Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο θέμα Ερασμός για όλους. ερασμός Plus. Ε, στην ημερήσια διάταξη βλέπετε ακόμη ε, για όλους. Έτσι, αυτό ήταν το όνομα το αρχικό της πρότασης της Κομισιόν και γι' αυτό το χρησιμοποιούμε για να ξέρουμε τι θα αλλάξουμε. Το Νοέμβριο του 2012 Είχαμε συζητήσει, είχαμε ψηφίσει για την έκθεση εδώ στην Επιτροπή και στη βάση αυτή δώσαμε εντολή στην ομάδα διαπραγμάτευσης για να προχωρήσει σε πραγματεύσεις με, με το Συμβούλιο. Ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής αυτής. Σκιώδης ήταν η Κατερίνα Νεμπιταλόβα, ο Μένα Ρατατού, η, Μακλάρ, η κυρία Μακλάρκιν και η κυρία Βεζιά. Συνεργάστηκα στενά με όλους τους σκιώδεις συζητητές για να βρούμε μια καλή συμβιβαστική λύση. Ξεκινήσαμε υπό Ιρλανδική Προεδρία. Πραγματοποιήθηκαν οι τριμερείς διάλογοι, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν στις 26 Ιουλίου. όταν η Κορεπέρ επιβεβαίωσε, ενέκρινε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων. Λάβαμε λοιπόν ε, ε, την τελευταία εβδομάδα μια επιστολή από τον κύριο Βεντσούνας. Νομίζω ότι έχετε λάβει την επιστολή αυτή. Στην επιστολή αυτή το Συμβούλιο λέει ότι θα εγκρίνει το κείμενο του Κοινοβουλίου αν το Κοινοβούλιο εγκρίνει το κείμενο σε πρώτη ανάγνωση. Αν δηλαδή την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο δεν υπάρξουν τροπολογίες, υπάρξει μια απλή ψηφοφορία δηλαδή, λόγω της πολύμινης διαπραγμάτευσης και λόγω της συμβαστικής λύσης την οποία έχουμε καταλήξει. Να πω για το έγγραφο αυτό ότι πρόκειται για μια εύλογη σύνοψη των ε, επιμέρους προγραμμάτων και ταυτόχρονα διατηρεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιμέρους τομέων. Όπως γνωρίζετε, έχετε λάβει, έχετε ενημερωθεί όλοι ότι δεν γίνεται να βάλουμε τα πάντα κάτω από μια ομπρέλα με τον τίτλο «Έρασμος για όλους», αλλά ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τους επιμέρους τομείς, Κομμένιους, Εράσμους, όλα αυτά είχαν ε, διαφορετικές ομάδες στις οποίες απευθύνονταν. Ακόμη και αν δεν, γνωρίζουν όλοι στην Ευρώπη τι είναι το κομμένιους, θεωρούμε ότι ήταν ε, σκόπιμο να διατηρηθούν αυτοί οι τίτλοι. Επομένως είμαστε ευτυχισμένοι που καταφέραμε να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και βεβαίως έχουμε το πρόγραμμα νεολαία σε δράση. Θεωρούμε ότι είναι πολύ θετικό το ότι διατηρήθηκε αυτό. Η επίσημη εκπαίδευση είναι εξίσου σημαντική με την ανεπίσημη και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μας. Το καλοκαίρι καταφέραμε να επιτύχουμε έναν ξεχωριστό προϋπολογισμό, τον λάβαμε μετά από πολύ μεγάλες προσπάθειες και ο συνάδελφος Μόκαγκάτ μας βοήθησε πολύ από την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Το πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα είναι για το 2014 στο 2020 και ο εξοπλισμός είναι ικανοποιητικός λάβαμε μια αύξηση του προπολογισμού κατά 47%. Δεν ξέρω, είναι ε, ε, μπορεί σε άλλου τομεί αυτό να μην θεωρείται ικανοποιητικό, αλλά για εμά αυτά τα 47% ε, είναι μια βελτίωση. Είναι τουλάχιστον 50% παραπάνω από την προηγούμενη. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε διάφορα με αυτήν την αύξηση. Έχουμε πλέον ένα δημοσιονομικό πλαίσιο 14,74 ε, ε, δισεκατομμυρίων ε, ευρώ. Στην Επιτροπή πολλές φορές είχαμε αντίθετη θέση με το Συμβούλιο και με την Κομισιόν, αλλά σε ένα ζήτημα είχαμε και εμείς διαφωνίες όσον αφορά τα μεταπτυχιακά και τα δάνεια Εκεί υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήθελαν πολλούς περιορισμούς. Στο τέλος όμως καταλήξαμε σε συμφωνία γιατί είπαμε ε, να μην διαθέσουμε ένα τόσο μεγάλο ποσό για το σκοπό αυτό και να το δούμε μετά τα, τα, τα πρώτα μισά χρόνια να το ξαναεξυλογήσουμε για να δούμε αν άξιζε εν τέλει τον κόπο να ε, διαθέσουμε τέτοιο ποσό για δάνεια για μεταπτυχιακά στο εξωτερικό. Συμφωνήσαμε επίσης διότι διαμορφώσαμε και την ε, επιστροφή των δανείων αυτών με, έναν, με, με περισσότερα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Δεν πρόκειται για τίποτα άλλο. Πρόκειται απλά για μια νέα προσφορά για όσου θα ήθελαν να την αξιοποιήσουν. Να ξαναευχαριστήσω λοιπόν όλου του σκιώδει συζητητέ και να ξαναπώ ότι πρόκειται πράγματι για μια καλή συμβαστική λύση που αποτελεί ξεκάθαρη πρόοδο σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Μεταξύ άλλων και επειδή έγινε πιο ευανάγνωστο το πρόγραμμα, πιο φιλικό προς το χρήστη. Τώρα μπορεί να βρει κανείς αυτά που ψάχνει. Στην αρχή εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να βρω αυτά που ήθελα να, να βρω, αλλά και αυτό το θέμα διευθετήθηκε. Να ξαναευχαριστήσω για άλλη μια φορά την Κομισιόν για την συνεργασία της. Ε, στο Συμβούλιο έχω το Συμβούλιο το έχω ευχαριστήσει ε, πολλές φορές. Είναι εδώ. Ναι, ωραία. Τότε χαίρομαι λοιπόν που είστε και οι δύο εδώ. Για άλλη μια φορά λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Και εύχομαι το πρόγραμμα αυτό να έχει την ε, επιτυχία που είχε και τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή να εξαντλήσουμε όλους τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Διότι είναι ένα από τα προγράμματα στα οποία δεν μένει ποτέ τίποτα. Ε, τίποτα ε, και είναι κρίμα γιατί τα τελευταία χρόνια ακούγαμε για το εράσμος δεν έχουμε λεφτά. Για το εράσμος πρέπει να έχουμε πάντοτε λεφτά. Όποιος ε, ενδεχομένως είχε άλλη άποψη θα πρέπει μάλλον να ψάξει αλλού. Θα ήθελε κάποιος άλλος κύριος από όσους συμμετείχαν στον τριμερή διάλογο να τοποθετηθεί, να πει κάτι. Όχι το ότι είναι όλοι επικαρμπημένοι μαζί μας, επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε στην ε, ψηφοφορία. Όποιος είναι... Συγγνώμη, αν κάποιος θέλει να πει κάτι, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Τόρις, πράγματι ε, επιτύχαμε κάποιες βελτιώσεις, αδιαμφισβήτητο αυτό, σε ό,τι αφορά και την αναγνωρισιμότητα των ε, επιμέρους υποπρογραμμάτων. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα εκ μέρους των Πρασίνων να πω ότι θα συμφωνήσουμε, θα ψηφίσουμε υπέρ του προγράμματος και εμείς διότι θεωρούμε ότι οι συμβαστικές λύσεις είναι σχετικά θετικές. Ωστόσο, έχουμε δύο σημεία κριτικής. Το ένα όσον αφορά τους, ε, την εμπλοκή των καταρτιζόμενων στο πρόγραμμα ε, Εράσμους και όσον αφορά την δημοσιονομική ε, στήριξη θεωρούμε ότι είναι μακριά από όσα ευχόμασταν αρχικά και θα εκφράσουμε αυτή την κριτική μας και στη συζήτηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να προσθέσω για άλλη μια φορά το πρόγραμμα Λεωνάρντο για τους καταρτιζόμενους δηλαδή δεν αυξήθηκε πολύ σε σχέση με το ε, παρελθόν, 25% διότι ένα μέρος αυτών που, έγιναν, ε, που γίνονταν παλιότερα ε, μέσω του προγράμματος αυτούς γίνονται πλέον μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αν δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, βεβαίω θα ζητούσαμε περισσότερα κονδύλια. Αλλά μα είπαν από την Κομισιόν και από το Συμβούλιο ότι όσα σχετίζονται με την ανεργία ε, εμπίπτουν στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και αυτή η τάση θα ενισχυθεί στο μέλλον. Στο μέλλον, κυρία να πω μόνο ότι τα κράτη-μέλη θα λάβουν υπόψη τους επιχειρησιακά ε, αυτές τις πτυχές σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Συμφωνώ και μπορώ να σας πω ότι στις ε, διαπραγματεύσεις για την ε, κυβέρνηση συνασπισμού θα επιμείνουμε να ληφθούν σοβαρά υπόψη όλα αυτά τα ζητήματα. Ξεκινώ λοιπόν την ψηφοφορία. Πέρας. υπέρ, Μαρίκε και εσύ υπέρ. Έχουμε λοιπόν 19 ε, συν 2 υπέρ, κανείς κατά, μία αποχή. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι κάναμε ένα πολύ σημαντικό και θετικό έργο. Προχωρούμε λοιπόν τώρα στο επόμενο σημείο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 Πάμε λοιπόν στην, ε, στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. 18 Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου η Επιτροπή Πολιτισμού συνέστησε μια ομάδα διαπραγματεύσεων για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα αυτό. Η συνάδελφος Σίλβια Κώστα ήταν η συγκήτριά μας. Ε, ήταν ο Ζωμαρί Κεμπέν, ο Κισάκ, Λότα Μπίσκι, ο Θανόν και ο Χάρμπλετ Πιντάλτσκι. Στον τριμερή διάλογο με την Ιρλανδική και τη Λιθουανική Προεδρία συνεργαστήκαμε στενά και στις 17 Σεπτεμβρίου του 2013 ε, καταλήξαμε σε συμφωνία. Θα ήθελα να δώσω το λόγο σύντομα στην Σίλβια Κώστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, δραστήρια συμμετοχή όλων, διότι οι διαπραγματεύσεις ήταν μακριές, ήταν σχηνοτενείς. Ευχαριστώ πολύ τους σκιώδεις, καθώς και τη γραμματεία για τη βοήθειά της και για την υπομονή που έδειξε. Νομίζω ότι με το πρόγραμμα αυτό το οποίο λαμβάνει υπόψη και τα οπτικοακουστικά μέσα για την Ευρώπη 2020 καθώς και τους ανθρώπινους ε, πόρους για την οικονομική ανάπτυξη και συνεργασία για την ευφύ ανάπτυξη. Νομίζω ότι με όλα αυτά κάναμε ένα θετικό βήμα προς το εμπρός. Και επειδή το ε, Κοινοβούλιο άκουσε όλους τους φορείς, τους συναδέλφους, τον ε, κόσμο των ε, οπτικοακουστικών μέσων της ΜΚΟ και, τον ε, πολιτιστικό, και το πολιτιστικό στερέωμα μπορέσαμε να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα δεδομένα καθώς και τους ειδικού στόχους και τα μέτρα που αφορούν τα μέσα και την, το συνολικό πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Λάβαμε υπόψη και ε, τον δανεισμό ο οποίος ε, προαπαιτείται και αποτιμήσαμε, αποτιμήσαμε τα υλικά και άειλα στοιχεία του πολιτιστικού στερεώματος καθώς και τον διαπολιτισμικό διάλογο και την κοινωνική συμμετοχή των νέων ιδιαίτερα και των επαγγελματιών. Θα ήθελα να πω ότι λυπάμαι, διότι παρά τις προσπάθειές μας έγινε περικοπή του προϋπολογισμού, έγινε περικοπή του προϋπολογισμού, αλλά μικρότερη από αυτή που αρχικά προβλέπαμε. Μιλάμε για μια στρατηγική επιλογή της Κομισιόν και σε σχέση με την προηγούμενη ε, επταετία ο προπολογισμός έχει περικοπεί κατά 10%. Συνεργαστήκαμε και με άλλες ε, επιτροπές και στον ορίζοντα 2020 και στα διαρθρωτικά ταμεία η λέξη πολιτισμός δεν είχε ενταχθεί και το τονίσαμε αυτό διότι μιλάμε για πολιτιστική κληρονομιά και στον ορίζοντα 2020 και στη, στα διαρθρωτικά ταμεία όπου δεν συμπεριλαμβανόταν. Μιλήσαμε και για τη συμμετοχή των διαρθρωτικών ταμείων στην διαδικασία ψηφιοποίησης μέσα στα πλαίσια των συνεργειών που δημιουργούνται για να προωθήσουμε τη δημιουργική αυτή Ευρώπη. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία της, ε, του Κοινοβουλίου έναντι της Επιτροπής. Αυτό καταδεικνύει μεγάλη αλληλεγγύη και συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι τηρήσαμε τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει, ιδιαίτερα ως προς τα οπτικοακουστικά μέσα και τους ανεξάρτητους φορείς που θα πλαισιώσουν τα ταμεία αυτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες και θα ήθελα να υποστηρίξετε αυτό το κείμενο που αποτελεί καρπό μιας μακροχρόνιας διαδικασίας. Σας ευχαριστώ Σίλβια. Στις 16 Οκτωβρίου ακούσαμε από τους επικεφαλής του Κόρεπερ. Λάβαμε επιστολή μάλλον, τον κύριο Βιτσιώνας, λάβαμε επιστολή με, που περίχε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, όπου ο πρέσβης επιβεβαιώνει ότι εάν ψηφίσουμε το κείμενο αυτό στο οποίο κατέληξαν σε συμφωνία τα τρία θεσμικά όργανα δεν θα αμφισβητηθεί πλέον και μπορούμε να θεωρήσουμε δεν θα υπάρξουν άλλες συνέχειες, αλλά θα εφαρμοστεί ως έχει. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι την Σίλβια καθώς και τους συζητητές. Δεν ήταν εύκολη δουλειά. να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό το business driven πρόγραμμα. Ο πολιτισμός ξεπερνά τα όρια αυτά. Ωστόσο και η Σίλβια μαζί με τους άλλους τα κατάφεραν καλά. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι. Και εγώ θα ήθελα να σχολιάσω από τη δική μας πλευρά. Επετύχαμε ορισμένες συμβαστικές λύσεις, να διορθωθεί δηλαδή η επιστημονική πορεία του προγράμματος, να υπάρχει περισσότερος χώρος για μη ε, κρατικές οργανώσεις και για μικρά προγράμματα. Η κριτική που ασκούμε στην ε, χρηματοδότηση είναι ότι δεν είναι επαρκής επιτύχαμε κάποια πρόοδο και γι' αυτό θα υπερψηφίσουμε το πρόγραμμα, ωστόσο διατηρούμε την κριτική μας και θα την καταστήσουμε και πάλι σαφή μέσα στα πλαίσια των συζητήσεων για το πολιετές οικονομικο πλαίσιο. Επειδή υπάρχουν πολλοί εδώ που παρακολουθούν παρατηρητές δηλαδή και τα δύο προγράμματα και ιδίω του πολιτισμού, δεν είναι εναρμονισμένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας δίνουν την δυνατότητα να προσθέσουμε μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε εθνικές δραστηριότητες. Δεν ασκούμε δηλαδή πολιτιστική πολιτική για την Γερμανία, τη Γαλλία ή την Εστονία. Προωθούμε κοινέ ιδέες σε μια προσπάθεια να τονίσουμε, να τονώσουμε και να προωθήσουμε την κοινή πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό επιδιώκουν τα προγράμματα αυτά. Άρα, δεν μπορούν να διατίθεται εκεί τα κονδύλια ύψους που διατίθεται στην ε, κοινή γεωργική πολιτική. Μόνο ευρωπαϊκά χρήματα κατευθύνονται στην γεωργική πολιτική και όχι εθνικά. Άρα, επειδή λένε μερικοί πώς είναι δυνατόν να δίνεται τόσα λεφτά στη γεωργία και τόσο λίγα στον πολιτισμό. Δεν μπορεί κανείς να τα συγκρίνει. Αφενός πρόκειται για μια καθαρά ευρωπαϊκή πολιτική, δηλαδή η κοινή γεωργική πολιτική και η άλλη πολιτική του πολιτισμού δηλαδή είναι προσθετική, είναι συμπληρωματική. Βεβαίως και θα μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερα κονδύλια, αλλά όπου δεν θέλει το Συμβούλιο, δεν θέλει. Έτσι λοιπόν εγώ είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που πετύχαμε έστω και μια αύξηση της τάξης του 8%. Υπάρχει άλλος κανείς που θα ήθελε να λάβει τον λόγο. Δεν βλέπω κανένα. Άρα προχωρούμε στην ψηφοφορία. Τέλος. Ψήφι Ανακοινώνω λοιπόν 20 συν 1, 21 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά και μία αποχή. Ευχαριστώ λοιπόν όλες και όλους. Τώρα μη μου φύγετε όλοι. Έχουμε να πούμε κάτι για το, για το βραβείο Λουξ. Μακλάκιν, μη φεύγετε. Είναι το δικό σου το βρετανικό φιλμ. Κάθε κάτω. Ε, λεπτά το βραβείο Λουξ. Παρακαλώ, μείνετε λίγο ακόμη. Πέντε λεπτά. Αρχίζουμε λοιπόν σήμερα αυτόν τον διαγωνισμό που είναι ο έβδομος στη σειρά του βραβείου Λουξ με τρία διαφορετικά, τρεις διαφορετικές ταινίες που προσφέρουν μια πραγματική ματιά σε πραγματικά ε, πολύ ενδιαφέροντα θέματα που βρίσκονται στην καρδιά των ευρωπαϊκών ιδιών και προβλημάτων. Για πρώτη φορά μάλιστα έχουμε και δύο ε, γυναίκες σκηνοθέτηδες. Αυτό μας προκαλεί μεγάλη περηφάνεια. Δεν το κάναμε επίτηδες, αλλά τι ωραία που έγινε έτσι. Και χαίρομαι επίσης που έχουμε και μια βρετανική ταινία στην, ε, στον διαγωνισμό και αυτό παρακα, σε παρακάλεσα εμένα να παραμείνεις. Λοιπόν, τρεις, τρεις ταινίες. Το ένα λέγεται «Μιέλε», Βαλέρια Γκολίνο είναι σκηνοθέτης και είναι Γάλλο-Ιταλική παραγωγή. Το δεύτερο, ο σπασμένος κύκλος ενός Βαν Γκρένιγκεν από το Βέλγιο και το τρίτο της Κρύο Μπανάρα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ταινίε αυτές ακούγονται και στην παγκόσμια σκηνή. Εμείς μάλιστα τι τις επιλέξαμε τις ταινίες αυτές πριν να το ξέρουμε, δηλαδή όχι εμεί αλλά η Επιτροπή, η Κριτική Επιτροπή. Υπάρχουν τώρα διάφοροι τρόποι να μπορέσει να παρακολουθήσει κανεί τι ταινίε αυτές. Από την 5η Νοεμβρίου και μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου έχετε τη δυνατότητα να δείτε τις ταινίε αυτές σε video on demand. Γράψτε ε, δύο λόγια στην γραμματεία του βραβείου Lux και ζητήστε τους ένα προσωπικό κωδικό ώστε να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τις ταινίες αυτές όπου θέλετε είτε στο σπίτι είτε εδώ χρειάζεστε πρόσβαση στο διαδίκτυο και τον κωδικό αυτό. Αυτές οι τρεις ταινίες μάλιστα έχουν υποτίτλους σε 24 γλώσσες. Μπορείτε να ζητήσετε λοιπόν την γλωσσική έκθεση που σας ενδιαφέρει. 24 γλώσσες. Πότε ξανά έγινε αυτό. Επίσης Τούτη την εβδομάδα στο κτίριο Μποζάρ θα γίνουν δύο ειδικές προβολές και στις 7 Νοεμβρίου, δηλαδή 7 Νοεμβρίου και στις 13. Όποιος θέλει δηλαδή μπορεί να πάει στο Μποζάρ σε ωραίο περιβάλλον και να παρακολουθήσει τις ταινίες αυτές. Επίσης όμως εδώ εντός του κτιρίου, δεν θυμούμαι τώρα από τι είναι, πότε αρχίζει η προβολή στον κινηματογράφο του τρίτου ορόφου, δεν ξέρει κανείς. Α, στις 25. Στις 25 ενδεκάτου αρχίζει η προβολή εκεί που είναι η Vox Box και μέχρι αρχών Δεκεμβρίου, δύο εβδομάδες. Μπορείτε εκεί να παρακολουθήσετε τις ταινίε και θα δείτε και στα φυλάδια πότε προβάλλονται οι ταινίε αυτές. Υπάρχει και κάτι ακόμη που είναι σημαντικό. Για κάθε ταινία λαμβάνετε στην γλώσσα σας μια περίληψη και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον αυτό έτσι ώστε να γνωρίζει κανείς εκ των προτέρων τι θα δει. Γι' αυτό και ευχαριστώ την ε, συνεργάτη μας Μαρισέλα και τον Ίγκριχ. Α, να, εκεί βρίσκονται. Του συγχαίρω λοιπόν γιατί έχει γίνει πραγματικά με θαυμάσιο τρόπο. Αυτές οι εβδομάδες προβολής των ταινιών πάνε πολύ καλά και σε άλλες χώρες της ε, Ένωσης. Στην Κολονία ήταν χθε η συνάδελφός μας την επόμενη εβδομάδα Μόναχο και Βερολίνο, όπου θα παραστώ και εγώ μαζί με άλλους συναδέλφους για να παρακολουθήσω τις δραστηριότητε αυτών των εβδομάδων προβολών. Α, σας τα δίνουμε και σε CD, άρα δεν χρειάζεται DVD, δηλαδή. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ε, ψάξετε στο διαδίκτυο. Τώρα, έγιναν και οι μερίδες κινηματογράφου στο Ζάγκρεμπ, επίσης στην Θεσσαλονίκη, όπου συμμετέχει η κυρία Παλιαδέλη στην Σεβίλη το Ευρωπαϊκό Film Festival. Εκεί προβάλλονται επίσης οι ταινίες. Στην Βιενάλε, στη Βιέννη, επίσης προβάλλονται οι τρεις αυτές ταινίες. Βρίσκω ότι είναι μια θαυμάσια ιδέα, αυτή η ιδέα που γεννήθηκε πριν από μια επταετία και η οποία μας έχει επιτρέψει στο μεταξύ να είμαστε παρούσες και παρόντες σε όλη την σκηνή των ε, κινηματογραφόφιλων, των συνεφίλ. Σε διάφορες πόλεις, στις Κάνες, στην Βενετία, στα διάφορα φεστιβάλ. Το βραβείο Λουξ λοιπόν υπάρχει, έχει μεγάλη ελκυστικότητα και δίνει τη δυνατότητα στις ε, ...αντιπροσωπήσει του Κοινοβουλίου στις διάφορες χώρες μέλη να προσεγγίσουν ανθρώπους που δεν θα τους έβρισκαν διαφορετικά. Διότι όταν μιλούν για γεωργική πολιτική ή βιομηχανική πολιτική, τότε προσέρχονται πάντοτε οι ίδιοι. Όμως όταν προβάλλονται ταινίε, τότε πάει όλος ο κόσμος που ενδιαφέρεται. Σε αυτές τις προβολές λοιπόν θα δοθεί και η δυνατότητα να μπορεί να ψηφίσει κανείς. Τα αποτελέσματα, μάλλον οι ψηφοφορίε αυτές δεν έχουν καμιά σχέση με τη δική μας ψηφοφορία που θα κάνουμε για να καταλήξουμε σε μια ταινία που θα νικήσει τον Δεκέμβρη. Αυτά τα βλέπετε και στα εγγραφά σας. Η ψηφοφορία αυτή που κάνουν οι θεατές και μπορούν να την κάνουν και μέσω διαδικτύου έχει τον σκοπό να διατηρήσει την επαφή με τους θεατές και μάλιστα μέχρι τον επόμενο χρόνο όπου θα προέρθουν οι νέες ταινίες από την ε, δράση της Κριτικής Επιτροπής. Και στην πόλη Κάρλο Βιβάρη θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και ορισμένους από αυτούς που συμμετέσχουν στην ψηφοφορία αυτή. Τα πρόσωπα αυτά να έχουν τη δυνατότητα λοιπόν να έρθουν να επισκεφθούν το Κάρλο Βιβάρη και να είναι παρόντες ή παρούσες στην, ε, στο φεστιβάλ. Άρα το βραβείο Λουξ ήδη έχει προσελκύσει τόσο ενδιαφέρον που δεν μας προβάλλει πλέον εμπόδια η Επιτροπή Προϋπολογισμών διότι αποδείχνεται ότι είναι ένα θαυμάσιο μέσο επικοινωνιακό και δημοσιότητας και μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τη δράση του Κοινοβουλίου με ένα νέο τρόπο. Επίσης στις 11 Δεκεμβρίου όταν θα απονεμηθεί το βραβείο εδώ στο Κοινοβούλιο θα έχουμε δηλαδή ψηφίσει, θα υπάρξει ένας νικητής, όλες οι ταινίες έχουν υποτιτλιστεί αυτό που θα νικήσει, δηλαδή η ταινία που θα νικήσει θα εκδοθεί και σε μια έκδοση για τυφλού. και στις 11 Δεκεμβρίου θα έχουμε λοιπόν μια διάσκεψη με τους δημοσιογράφους και παρακαλώ βρείτε χρόνο να έρθετε διότι θα προσκαλέσουμε προσωπικότητες μεγάλου κύρους από τον χώρο του κινηματογράφου. Θα έχουμε τον επικεφαλής της Biennale της Βενετίας, Επίση την ε, επικεφαλής του Άρτε που μας συνοδεύει σε όλη αυτή την προσπάθεια του βραβείου Λουξ. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να εμφανίσουμε το κοινοβούλιο και να δώσουμε μια εικόνα, μια εντύπωση που δεν έχει κανείς διαφορετικά. Αυτό δεν σημαίνει διόλου ότι σπαταλούμε τα χρήματά μας. Χρησιμοποιούμε τα κονδύλια της επικοινωνίας για να φέρουμε τους ανθρώπους σε επαφή με ταινίε και με θέματα τα οποία κάποια στιγμή άπτονται και των εργασιών μας. Η ταινία Welcome για τους Γάλλους ήταν για το άσυλο ή η ξένη επίσης που κέρδισε το βραβείο. Φόνη λόγω τιμής ήταν το αντικείμενό της. Αυτές οι ταινίες λοιπόν είναι πραγματικά εξαιρετικές και μας δίνουν τη δυνατότητα να προκαλέσουμε τη συνειδητοποίηση του κόσμου για προβλήματα που σημειώνεται και σε όλη την Ένωση. Να, βλέπετε εδώ τώρα τα τρία φυλάδια, όπου να δείτε τα σχετικά. Βλέπετε και το DVD που λαμβάνετε μόνο όσοι είστε παρόντε και παρουσε εδώ οι άλλοι, τόσο το χειρότερο για αυτούς. Μπορείτε να ζητήσετε βέβαια το DVD ή να το βρείτε όπως είπα το film σε video on demand. Αυτά ήθελα να πω για το θέμα του βραβείου Lux. Επίσης κάθε χρόνο όταν παρουσιάζουμε την ταινία για πρώτη φορά στην Βενετία, δηλαδή τις τρεις προτινόμενες υποψήφιες ταινίες, μαζί με το Europa Cinema προσκαλούμε 28 νέους ανθρώπους από τις 28 χώρες μέλη, κινηματογραφόφιλους, όχι σκηνοθέτες κτλ. Μπορεί να είναι σπουδαστές, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Προσέρχονται τα πρόσωπα αυτά και μένουν στη Βενετία όλοι μαζί, παρακολουθούν όλες τις ταινίες στην πιενάλε, μπορούν να συνομιλήσουν, μπορούν να φτιάξουν φιλίες. 28. Πού αλλού θα, βρείτε, θα βρείτε 28 νέους όλων των εθνικοτήτων για να μπορέσουν να συζητήσουν και να συνάψουν φιλικές σχέσεις. Και για πρώτη φορά ήταν φέτος και οι Κροάτες. Άρα δίνουμε μια δυνατότητα σε αυτούς τους νέους. Αυτοί ασχολούνται με τα blog και έχουν κάνει και μικρές ταινίες ενός λεπτού. Κάθε φορά που θα προβάλλεται μια ταινία θα προβάλλουμε και αυτές τις μικρές ταινίες των ε, νέων των νεαρών ε, αυτών, γιατί δίνει και μια μυρωδιά για τα πράγματα που ε, παράγουν και τι προκύπτει από αυτή τη συνάντησή τους. Πήγα και στην Πιενάλε προδιετία στο Βερολίνο και Ήρθε λοιπόν ένας νεαρός και με σκούτησε και μου λέει στα αγγλικά είστε η κυρία Πακ και μου λέει είμαι ένας από τι 27. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μου είπε ο νέος εκείνος ότι ήταν τέσσερις στην Βιενάλε ε, ορισμένοι είχαν έρθει με auto-stop, άλλοι Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε στα χέρια μας ένα θαυμάσιο εργαλείο και γι' αυτό θα θυμίσω και ποιος ήταν αυτός που επινόησε αυτή τη θαυμάσια ιδέα, ο κύριος Ονεστά, των πράσινων. Βεβαίως είχε και την υποστήριξη και άλλων, γιατί ίσως χρειάζεται και κάπως μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα. Την είχε και γι' αυτό καταφέραμε να διατηρήσουμε αυτή τη θαυμάσια υπόθεση ήδη μια επταετία. Λοιπόν, καλή διασκέδαση. Ζητήστε και το βίντεο on demand και για τα γραφεία σας αν θέλετε. Τώρα, το λόγο. Μπόρις, Πιέτρο. Ευχαριστώ. Ήθελα να ευχαριστήσω που έχετε στηρίξει τόσο πολύ το βραβείο. Εγώ έχω συμμετάσχει και σε εκθέσεις για τον κινηματογράφο και στη Γερμανία και στην Πολωνία βλέπω ότι τα γραφεία πληροφοριών του Κοινοβουλίου κάνουν τρομερή promotion για τις ταινίες αυτές. Εγώ βρέθηκα μαζί με νεαρούς και νεαρές στις προβολές των ταινιών αυτών και είδα ότι συζητούν τα προβλήματα της Ευρώπης. Αυτή η προσπάθεια αξίζει να ενισχυθεί και αυτές οι ορθές πρακτικές που γίνονται ήδη στη Γερμανία, στην Πολωνία, που τις διεξάγουν τα γραφεία πληροφοριών του Κοινοβουλίου μας, που στηρίζουν και προωθούν τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και την ευρωπαϊκή ταινία, όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά. Μπορούν να επιτευθούν μέσω των ταινιών. Και ελπίζω του χρόνου να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο προσπάθεια αυτή. Ανρή Καβαντά. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω μία πληροφορία προς εσάς και όλους τους συναδέλφους. Στα πλαίσια του βραβείου Λούξε στη Γαλλία, το ευρωπαϊκό, ε, γαλλικό, ευρωπαϊκής ε, γαλλικό κείμενο ε, προωθεί αυτό το κίνημα που είναι μία ΜΚΟ, αποφάσισε σε 20 γαλλικές ε, πόλεις να προωθήσει όλα τα βραβεία Λουξ μέχρι τώρα, εάν ε, επιτραπεί στη Λίλη, καν στο Μπορντό, Μομπελιέ και άλλες ε, πόλεις, δηλαδή να προβληθούν όλα τα έργα των μέχρι τώρα, του μέχρι τώρα βραβείου Λουξ δωρεάν στις γαλλικές αυτές πόλεις για να δούμε τα ευρωπαϊκά θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα τους σκηνοθέτες αυτούς. Η Σίλβια. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τόρι Σπάκ για τη δέσμευσή της και το πάθος που καταδεικνύει στη Βενετία και στο Κάρλο Βιβάρι. Είδαμε ότι προωθούνται αυτές οι πρωτοβουλίες πολύ κινηματογραφόφιλοι συμμετέχουν σε αυτές τις ε, προβολές. Έχουμε 28 νέους ανθρώπους που προσέρχονται και προβάλλουν ε, ε, τις θέσεις αυτές του συνομήλικους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει η καινοτομία από πέρσι, να προωθήσουμε δηλαδή αυτά τα φεστιβάλ και στη Ρώμη τους επόμενους μήνες θα προβληθούν ε, έργα στο Μάξι καθώς και στο σπίτι του κινηματογράφου της ε, Ρώμης. Υπάρχει μεγάλη, υπάρχουν πολλαπλά αιτήματα προς αυτή την κατεύθυνση και δεσμευόμαστε όλοι. Η Σίλβια ήταν πάντα μαζί μου όταν ήμασταν στην Βενετία, γιατί το συζητάμε αυτό με τους ε, νέους και ιδιαίτερα εκείνους που ζουν κοντά στη Βενετία και μπορέσαν να προσέλθουν. Αυτό ήταν κάτι το εξαιρετικό, κυρία Χάνιμπαλ. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για τον ενθουσιασμό σας, διότι συμμετέχει και ένα βρετανικό έργο στο διαγωνισμό αυτό. Είδα τις πληροφορίες ε, για αυτό το έργο και νομίζω ότι είναι πολύ καυστικό και εγώ είμαι ιδιαίτερα ενθουσιώδης. Όπως είπατε, το έργο αυτό αντικατοπτρίζει τα κοινωνικά προβλήματα που υφίστανται και αυτό, είναι, αυτό αποτελεί και τη δύναμη του βραβείου Λουξ. Δηλαδή έχουμε μία διαφορετική παρουσίαση των πραγμάτων. Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιώδης φέτος και να συγχαρώ όλους όσους συμμετείχαν. Ευχαριστώ. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τα όσα εξήγησε η Doris Πακ και η διοργάνωση χθε στην κολονία ήταν υπέροχη. Ήταν πραγματικά πληρέστατη η αίθουσα του κινηματογράφου και τρει ταινίε, η μια μετά την άλλη, μέσα σε μια μέρα. Πραγματικά είναι και σκληρή δουλειά να τις παρακολουθήσει κανείς και δεν είναι και εύκολα φιλμ αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν πραγματικά θαυμάσια εκδήλωση. Χθες είχα και την ευκαιρία και τη χαρά να γνωρίσω ένα εκπρόσωπο της ε, ε, Κριτικής Επιτροπής όλες τις ε, τελευταίες περιπτώσεις ήταν θαυμάσεις ταινίε και καταλήγουμε έτσι να μπορούμε να επιρρέψουμε σε επαφή με ανθρώπους που δεν φτάνουμε να τους πλησιάσουμε με πολιτικές συζητήσεις. Δεν, δεν είναι απαραίτητο οι ευρωπαϊκέ ταινίε να φορτώνονται πάντοτε όλα τα βάρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή του κόσμου. Είπα λοιπόν στην ε, εκπροσώπηση χθε τη Κριτική Επιτροπή, διαλέξτε μια ωραία έξυπνη, χαριτωμένη ευρωπαϊκή κομμωδία. Νομίζω ότι θα μπορέσει να παρουσιάσει και ίσω μάλιστα να προσεγγίσουμε ακόμα περισσότερου ανθρώπου από το να επιλέγουμε πάντα ταινίε που είναι αργέ, έχουν αργού ρυθμού και είναι και πάρα πολύ φορτωμένε. Εάν καταφέρουμε οι άνθρωποι να φύγουν χαρούμενοι, πετώντα από τον κινηματογραφό και όχι έτσι με ένα βάρο, ίσω να είναι ακόμα καλύτερα. Τα είπα αυτά λοιπόν στον εκπρόσωπο τη Κριτικής Επιτροπή. εχθές και ελπίζω να βοηθήσει. Ωραία θα ήταν του χρόνου να ε, βραβεύσουμε μια κομμωδία. Ε, Doris δεν μπορεί να φανταστεί πόσε φορέ το έχω πει στο μέλο αυτό τη Κριτικής Επιτροπή έρχονται συνάδελφοι και μου λένε μα είναι τόσο θλιμμένες οι ταινίες αυτές. Ναι βεβαίως ο κόσμος δεν είναι ε, μόνο χαρούμενος. Αλλά η Οσονολή αυτή η ταινία δεν ήταν μόνο θλιμμένη, ήταν και χαρούμενη και ρομαντική. Τέλος πάντων, έχω για ορισμένους Γερμανούς άνδρες τουλάχιστον την αίσθηση ότι περισσότερο αυτό τους αρέσει. Τα είπα και εγώ αυτά. Όμω εμεί δεν είμαστε στην Κριτική Επιτροπή και στην Κριτική Επιτροπή πρέπει να προσέχει κανεί διότι ορισμένοι θέλουν ένα κινηματογράφο δύσκολο και απαιτητικό. Εγώ μιλώ βεβαίω συνεχώ με τα μέλη τη Κριτική Επιτροπή αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Σε αυτέ τι τρει ταινίε πάντω περιλαμβάνεται μία όπου θα σα κάνει να γελάσετε πολύ αν και δεν είναι εντελώ απροβλημάτιστη, μπορεί όμω να γεράσει κανεί ε, με αυτά που βλέπει στην ταινία. Τέλο πάντων, αυτά. Ναι, Πιέρ. Α, ο Ζαμαρή. Υπήρχε μια πολύ ωραία κομμωδία ε, του Φρεντερίκ Κλαπής που λεγόταν ο Μπέρζ Εσπανιόλ που δεν έλαβε το βραβείο αλλά δεν πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι δηλαδή μπορούμε να βγάλουμε το μαντιλάκι μας και να κλάψουμε αλλά μπορούμε να είμαστε και ευτυχείς υπάρχουν δύο χρήσεις Είχαμε και το έργο, το, ένα άλλο έργο, το Κιλιμαντζάρο, που ήταν πολύ ωραίο και γελάσαμε και κλάψαμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αλλά υπάρχουν συνάδελφοι που δεν, τα, δεν το λαμβάνουν υπόψη, θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι πιο ε, αισιόδοξα τα έργα. Σίγουρα Μαρισέλα και εσύ Ένριχ. Αυτή είναι αυτά τα δύο πρόσωπα που έκαναν όλη τη δουλειά μόνοι τους. Είναι καταπληκτικοί και εργάστηκαν σκληρά πραγματικά μέχρι πολύ αργά τη νύχτα. Θαυμάσια. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Θεματικό τμήμα Β, ποιότητα στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Έχουμε τον ερευνητή μας, τον κύριο Γκέρτιαν Λίντεμπον, είναι σύμβουλος στην Παντέια. Τον Μάιο του 2011 το Κοινοβούλιο θέτησε την έκθεση Hannibal για την ε, προσχολική μάθηση. Σκόπος ήταν η καλύτερη εξέλιξη της μάθησης στα πρώτα προσχολικά χρόνια. Προσπαθήσαμε να διεξαγάγουμε μια έρευνα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Την προηγούμενη χρονιά λοιπόν η μονάδα μας ανέθεσε την διεξαγωγή ε, μελέτης και σήμερα έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Γκέρτιαν Λίντεμπομ Κύριε Λίντεμπομ, σας παρακαλώ. 15 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας, το ανώτατο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τα ευρήματα της μελέτης μας εδώ στην Επιτροπή σας. Ε, η μελέτη αυτή διεξήχθη από μένα και τους συναδέλφους μου στην Παντέια. Ε, θα ήθελα να σας ε, πω για το ιστορικό, για τον στόχο της μελέτης, για το πλαίσιο εξελόγηση, τις, τα κύρια ευρήματα, τα συμπεράσματα, τις ε, συστάσεις και τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω κάποια πράγματα για το υπόβαθρο αυτής της μελέτης. Φυσικά οι πολιτικές για την ΠΕΦ ε, επηρεάζουν όλους τους γονείς ε, αρχικά ε, αποσκοπούσαν στην εμπλοκή περισσότερο των γυναικών στην αγορά εργασίας. Αλλά όλο και περισσότερο ε, στόχος είναι να δοθούν ίσες ευκαιρίες στα παιδιά για την ε, ανάπτυξή τους. Έτσι λοιπόν έχουμε μια μεταβίβαση πολιτική, μια μετάβαση πολιτικής τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Από, τα, από περισσότερες θέσεις προσχολικής εκπαίδευσης σε καλύτερες στην ε, ανακοίνωσή της ε, η Κομισιόν το 2011 είπε ότι η ΠΕΦ είναι θεμελιώδης για την επιτυχημένη διαβίου μάθηση, την κοινωνική ένταξη, την προσωπική ανάπτυξη και την απασχολησιμότητα σε ε, επόμενο στάδιο. Ω συνέχεια στους στόχους της Βαρκελόνης και της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 ε, τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να δημιουργηθούν 90%, για 90% των παιδιών από ηλικίες άνω των τριών ε, θέσεις προσχολικής εκπαίδευσης. Αντιστοίχως ε, η Κομισιόν έκανε βήματα στον ορισμό της ποιότητας. Ποια είναι λοιπόν ε, η πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 2002 στην Βαρκελόνη τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να ε, δημιουργηθούν, να εξασφαλιστούν ε, για το 90% των παιδιών άνω των τριών ετών θέσεις πλήρου πλήρους ε, προσχολικής εκπαίδευσης και 33% για τα παιδιά από 0 έως 2 ετών. Ωστόσο, ε, οι στόχοι αυτοί δεν έθεταν καμία ποιοτική ε, πτυχή, ενώ η νομοθεσία ορίζει ρητά ότι η ορθή ανάπτυξη πρέπει να συνοδεύεται, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της ε, ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης. Το 2011 η Κομισιόν και το ε, Κοινοβούλιο καθόρισαν περισσότερα ποιοτικά στοιχεία όσον αφορά την ε, ΠΕΦ ως κατευθυντήριε γραμμές για τα κράτη-μέλη. Ωστόσο, ε, αν κοιτάξουμε πιο κοντά, τα, ε, πιο διεξοδικά τα κράτη-μέλη, μπορούμε να βρούμε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Για να απαντήσουμε ε, εξετάσαμε, μια, χρησιμοποίησαμε μια προσέγγιση διπλή. Κοιτάξαμε αφενός τις ε, εξελίξεις όσον αφορά την ΠΕΦ σε ε, ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών. Προσπαθήσαμε λοιπόν να ε, συνεκτιμήσουμε μελέτες που υπάρχουν. Συγκεκριμένα επιλέξαμε ε, έξι χώρες και κάναμε συνεντεύξεις με, με ενδιαφερόμενα μέρη, αναλύσαμε. Συγκεκριμένα οι ε, χώρες που επιλέξαμε ήταν η Ισπανία, οι κάτω χώρες, η Ρουμανία, η Ιρλανδία, η Γερμανία, η Βόρεια Ιρλανδία, η Βεσφαλή και η Φιλανδία. Η μελέτη αυτή έγινε με σκοπό να καλυφθούν και διάφορες ε, παιδαγωγικές μέθοδοι και κουλτούρες. Θέλαμε να μάθουμε ε, τι συμβαίνει κάτω, στη βάση. Γιατί πολλές φορές ε, υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Η έρευνά μας διαπίστωσε ότι υπάρχουν πολλές καλές πρακτικές οι οποίες περιγράφονται λεπτομερώς σε όλη την έκθεσή μας. Καθώς μιλούμε, η Κομισιόν εφαρμόζει μια ανοιχτή μέθοδο συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών για να ε, καθορίσουμε ένα πλαίσιο. Επειδή ακόμα βρισκόμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο, βασίσαμε την προσέγγιση μας για, στις ε, προτεραιότητες ε, που βλέπουμε που υπάρχουν τόσο στο έγγραφο της Κομισιόν όσο και ε, στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Βλέπετε εδώ στον πίνικα... ότι ε, συγκρίναμε τις προτεραιότητες της Κομισιόν και εκείνες του Κοινοβουλίου. Ε, κατά γενική ομολογία καλύπτουν παρόμοια θέματα. Και μετά είδαμε και εξετάσαμε και τα κράτη-μέλη. Είδαμε την πρόσβαση, τα πολιτικά νομικά οικονομικά πλαίσια, το προσωπικό, τα αναλυτικά προγράμματα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τέλος ε, πώς ε, σχεδιάζεται η εμπλοκή των γονέων. Αυτά ήταν η, τα, τα, τα σημαντικότερα ε, σημεία προσοχής της μελέτης μας. Τα κυριότερα ευρήματα μας. Ο στόχος 95% συμμετοχής είναι ο μοναδικός που ορίζεται ρητά. Βλέπετε εδώ με μπλε χρώμα τα αποτελέσματα. Να σας πω ε, κάποια πράγματα για, τα, για τον πίνακα που βλέπετε στην οθόνη. Ε, εμφανίζεται λοιπόν η ε, εμπλοκή μεταξύ, ε, η συμμετοχή μεταξύ 2000-2010 για τα παιδιά άνω των 4 ε, ετών με κίτρινο βλέπετε τις διαφορές που έχουν γίνει από το 2000 και έτσι έχουμε το, ε, συνολικά το επίπεδο του 2010. Με κόκκινο βλέπετε ότι υπάρχει μια συμμετοχή όπου υπάρχει ε, μείωση της συμμετοχής. Βλέπετε ότι υπάρχει μια σαφή στάση αν και υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές βεβαίως ταυτόχρονα μεταξύ των κρατών μελών αν συγκρίνει κανείς ε, τα επίπεδα του 2000 με, με εκείνα του 2010 με πολύ μικρές μειώσεις. Ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας βεβαίως και την ε, δυνητική επίπτωση της ε, οικονομικής κρίσης από το 2008. Έχουμε σαφείς ενδείξεις ότι η κρίση αυτή είχε αρνητικές επιπτώσεις στην ε, ΠΕΦ και αυτά ενδεχομένως ακόμη να μην έχουν καλυφθεί πλήρως, οι επιπτώσεις αυτές να μην έχουν καλυφθεί πλήρως από την μελέτη. Άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους, έχασαν εισόδημα, ταυτόχρονα οι κυβερνήσεις ε, περικόπτουν ε, την ενίσχυση. Γι' αυτό πολλοί γονείς επιλέγουν να προσέχουν τα παιδιά τους οι ίδιοι. Αυτό θα πρέπει να το, έχουμε, ε, να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια. Επίσης όμως υπάρχει και ένας σημαντικός κίνδυνος. Αφενός ε, υπάρχει ο, ο κίνδυνος τα κράτη-μέλη να εστιάσουν μόνο στις δαπάνες και όχι στην ποιότητα. Επίσης, ε, πολλές φορές οι προσπάθειες κατευθύνονται στις ομάδες που είναι εύκολο, εύκολα προσβάσιμες, ενώ αυτές που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες θα ήταν εκείνες που θα ωφελούνταν περισσότερο. Βλέπετε εδώ την ε, ε, Φιλανδία που έχει το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής. Ε, στη Φιλανδία γίνονται προσπάθειες ώστε και ομάδες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση κοινωνική έχουν πρόσβαση στην ΠΕΦ. Στόχος λοιπόν θα, θα ήταν να διευρυνθεί και όχι απλά να ε, αυξηθεί η συμμετοχή. Οι πολιτικές προσχολικής εκπαίδευσης θα έπρεπε να είναι πιο περιεκτικές, να απευθύνονται σε περισσότερες ομάδες και όχι απλά να έχουν στόχο την αύξηση των, ε, των αριθμών συμμετοχής. Σχεδιασμός ένα άλλο στοιχείο. Σύμφωνα με τις μελέτες που έχουμε στη διάθεσή μας, είναι καλύτερο να έχουμε ε, ενιαοποίηση των διαφόρων ε, υποσυστημάτων. Υπάρχει λοιπόν ε, μια τέτοια σαφή στάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην, ε, σε πολλές ευρωπαϊκές ε, χώρες υπάρχει ακόμα μια πολύ ισχυρή διαχωριστική γραμμή μεταξύ της ε, προσχολικής φροντίδας και στα τρία χρόνια της ηλικία και στο επόμενο στάδιο. Η, ποιο... η διασφάλιση ποιότητας τώρα ε, πολλές φορές απευθύνεται στοχεύει στην ε, κατάρτιση ελάχιστων ε, προτύπων. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους παρόχους προσχολικής εκπαίδευσης να κάνουν περισσότερα από ό,τι ε, ορίζεται από την νομοθεσία. Καλό παράδειγμα, για παράδειγμα βρήκαμε στην Ιρλανδία, όπου υπάρχει ένα πλαίσιο εθνικής ποιότητας, Σιέλτα το οποίο ενθαρρύνει τους ε, καθηγητές να διευρύνουν και να προωθούν την ποιότητα και όχι απλώς να τηρούν τα ελάχιστα πρότυπα. Ενθαρρύνονται επίσης να ανταλλάσσουν γνώμες με τους συναδέλφους τους ώστε να προωθούνται και να βελτιώνονται διαρκώς τα πρότυπα. Ωστόσο, ε, τέτοιες πρωτοβουλίες εξαρτώνται πάντοτε από τη χρηματοδότηση. οι δαπάνες, τα κονδύλια που έχουν στη, στην διάθεσή τους, ε, που διατίθενται μάλλον για την προσχολική εκπαίδευση, βρίσκονται υποπίεση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχετίζεται βεβαίως και με την ε, κρίση. Μπορούμε, ε, διαπιστώσαμε μια θετική σχέση μεταξύ των δαπανών και της ποιότητας και αυτό αντανακλάται και στη στην βαθμολογία ε, πίζα. Τώρα για το προσωπικό, τα προγράμματα και την εμπλοκή των γονέων. Στις έξι χώρες ε, διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά ότι υπάρχει ανάγκη ελάχιστων προσόντων Θα πρέπει διαρκώς να ελέγχεται η επίδραση με τα παιδιά και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό το προσωπικό να έχει αυτές τις ικανότητες. Υπάρχουν βεβαίως ε, ε διάφορα, διάφο, διάφορες ελάχιστες απαιτήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ με διάφορα χρώματα μπορείτε να βρείτε ε, τις ελάχιστες απαιτήσει για να εργαστεί κανείς στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι ε, ενισχύονται όλο και, περισσότερα, ε, όλο και περισσότερο τα επαγγελματικά κριτήρια στην ε, Βόρεια Ιρανία Βεστιφαλία... υπήρχαν άτυπες δομές προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας και εκεί διαπιστώσαμε ότι οι εργαζόμενοι σε, αυτούς, σε αυτές τις δομές ε, προσπαθούσαν να βελτιώσουν τα επαγγελματικό τους, τα επαγγελματικό τους προσόντα. Γενικά, εν πάση περιπτώσει, βρήκαμε ότι υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη μεγαλύτερη εστίαση στην εκπαίδευση. Και αυτή η τάση αφορά και την προσχολική εκπαίδευση. Η η... Επίσης υπάρχει ε, πολλές χώρες που εισάγουν έτος υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, Ρουμανία, Φιλανδία. Τώρα όσον αφορά τον ε, ρόλο των γονέων, πάλι υπάρχουν πολλές ε, διαφορετικές ε, πολιτικές αλλά πάντως αναγνωρίζεται ο ρόλος των γονέων. Τώρα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι εξελίξεις πολιτικής για την ΠΕΦ βρίσκονται ακόμη σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης παρότι έχουν ε, ε, τεθεί στόχοι όσον αφορά τη συμμετοχή των νέων παιδιών, δεν υπάρχει κοινή αντίληψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών για το τι ακριβώς συνιστά ποιότητα στην προσχολική εκπαίδευση. Στη βάση των ε, διαφορετικών στοιχείων της ποιότητας που εξετάσαμε, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία, αλλά και διαφορά γνωμών, απόψεων για το τι είναι οι ορθές οι βέλτιστες πρακτικές. Κάποιες χώρες έχουν ε, συγχωνευμένα συστήματα ΠΕΦ, ενώ άλλα έχουν διαχωρισμένα συστήματα. Υπάρχουν ε, κάποιες χώρες καταρτίζουν κεντρικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα, άλλες το αφήνουν στους παρόχους. Είναι σημαντικό οι πολιτικές που θέτουν ποσοτικούς στόχους να μην αγνοούν τις ομάδες που είναι δύσκολο να ε, έχει πρόσβαση κανείς. Στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση κανείς. Στόχος είναι να συμβιβάσουμε τις διαφορετικές πολιτικές και προσεγγίσεις Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αποκτήσουμε δηλαδή μια κοινή αντίληψη για το τι είναι η ΠΕΦ. Ποιε είναι λοιπόν οι συστάσεις για να προωθήσουμε περισσότερο αυτό το ε, ποιοτικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακριβώς επειδή βρισκόμαστε αυτό, σε αυτό το πρώιμο στάδιο, τα θεσμικά όργανα μπορούν να δημιουργήσουν ένα πολιτικό πλαίσιο στο οποίο θα μπορέσουν τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τις πολιτικές τους. Έτσι, ε, για το σκοπό αυτό ορίσαμε κάποιους ε, κρίσιμους παράγοντες ε, ανοιχτής μεθόδου συντονισμού. Οι παράγοντες αυτοί, όπως βλέπετε, είναι ε, η πολιτική συμμετοχή, η ευαισθητοποίηση, οι δομές, η, θέσπιση σαφών στόχων και δικτών, η εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών και ε, η αξιοποίηση των, ε, της πυκλομορφίας για να προχωρήσουμε μπροστά. Θα το εξηγήσω λίγο καλύτερα για να σας πω πώς μπορούμε να ε, το Κοινοβούλιο να λάβει βήματα ώστε να ενθαρρύνει την Κομισιόν να προχωρήσει στα απαραίτητα μέτρα. Πρώτα, να ε, προωθήσουμε την πολιτική ε, συμμετοχή, την πολιτική εμπλοκή. Αν κάτι δεν είναι ενδιαφέρον για τους πολίτες, ε, τότε η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού μάλλον δεν θα είναι επιτυχημένη. Πολλά κράτη-μέλη έχουν λάβει βήματα για την βελτίωση της ποιότητας και της διαθεσιμότητας της ΠΕΦ. Από αυτή την άποψη λοιπόν η πολιτική εμπλοκή φαίνεται ότι είναι ικανοποιητική. Ωστόσο, ε, αυτή τη στιγμή η ποιοτική ΠΕΦ ε, είναι μια ανησυχία για τα κράτη-μέλη, για πολλά κράτη-μέλη, αλλά όχι για όλα. Οι πολιτικές στον τομέα αυτό ε, είναι σχεδόν αποκλειστικά εθνικές. Δεν υπάρχει πλαίσιο ευρωπαϊκό μέσω του οποίου να, ε, να μπορούν να συγκριθούν οι πολιτικές. Αυτή τη στιγμή ε, καταρτίζεται ένα γλωσσάριο από την Κομισιόν για την ορολογία που χρησιμοποιείται και αυτό το γλωσσάριο θα μας βοηθήσει στις ε, μελλοντικές συζητήσεις μας για το ζήτημα αυτό. Συνιστούμε το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν να μην υποτιμήσουν ε, αυτή τη διάσταση της κοινή αντίληψης και της κοινή ορολογίας. Επίσης, χρειάζεται μια θεσμική υποστήριξη για να έχουμε επιτυχημένη ε, ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Αυτή τη στιγμή η θεματική ομάδα ε, εργασίας ε, ε, έχει ήδη συσταθεί. Επίσης υπάρχει συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Από αυτή την άποψη ε, υπάρχουν θεσμικά όργανα για συντονισμό. Τέταρτον, απαιτούνται σαφείς στόχοι, δείκτες, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να διαπιστώνουν την πρόοδο που κάνουν σε σύγκριση με άλλα κράτη-μέλη. Κανένα κράτος μέλος ε, προφανώς δεν θα ήθελε να ε, είναι τελευταίο σε μια τέτοια ανάλυση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο στόχος 95% συμμετοχής για παιδιά άνω των 4 ετών. Ωστόσο, όπως είπα και νωρίτερα, αυτός ο στόχος ε, μας οδηγεί πολλές φορές στη δημιουργία περισσότερων και όχι απαραίτητα καλύτερων θέσεων προσχολικής εκπαίδευσης. Άρα πρέπει να δημιουργηθούν και ποιοτικοί δείκτες. Και τα ευρωπαϊκά όργανα θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους πολύ σοβαρά αυτά, γιατί και αυτά θα επηρεάσουν σημαντικά την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Όπως είπα, ε, είναι σημαντικό να έχουμε συγκεκριμένους στόχους και δείκτες για την προσχολική εκπαίδευση σε όλη την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών. Επίσης, κρίσιμο ζήτημα. Θα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση από τα κάτω προς τα πάνω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομάδα ενδιαφερόμενων μερών, αλλά πάντως αυτή δεν έρχεται σε επαφή με την θεματική ομάδα εργασίας. Είναι σημαντικό σε κάποιο σημείο, σε κάποιο στάδιο η Κομισιόν να εμπλέξει τα ενδιαφερόμενα μέρη και να τα φέρει σε επαφή με τη θεματική ομάδα. Η, η καθοδήγηση σε, ευρωπαϊκή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να είναι βιώσιμη, να είναι επιτυχημένη μόνο ε, αν ε, ακούγονται και οι γνώμες των ενδιαφερόμενων μερών. Τέλος, αν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ κρατών μελών αν υπάρχει κάποιο κράτος μέλος που δεν, δεν έχει διάθεση να αναλάβει δράση, μπορούν τα ίδια τα κράτη-μέλη να αναλάβουν το στόχο να ενθαρρυνθούν, να ενθαρρυνθεί η κατάρτιση τέτοιων πολιτικών. Αυτή τη στιγμή ε, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τις, συγκρούσεις, τις ενδεχόμενες συγκρούσεις μεταξύ των κρατών μελών. Πάντως οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών μπορούν να μας οδηγήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο. Μέσω της Μέσω των συστάσεων αυτών, η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο μπορούν να υποστηρίξουν την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού για να ενισχυθεί η ποιοτική ΠΕΦ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι μπορούν να κάνουν τώρα τα κράτη-μέλη για την προώθηση της ποιότητας Συνοψίζοντας, να σας πω τα κυριότερα σημεία που ε, εντοπίσαμε σε επίπεδο κρατών μελών. Πρώτα απ' όλα, είναι απολύτως απαραίτητο οι πολιτικές στα κράτη-μέλη να βασίζονται στις ενδείξεις. Πολλές φορές βρήκαμε ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται δεν είναι αρκετά τεκμηριωμένες. Πολλές ε, βασίζονται σε αμερικανικές ε, μελέτες και ενώ δεν υπάρχουν ανάλογες ευρωπαϊκές μελέτες μεγάλου εύρους. Επίσης δεν δίνεται ιδιαίτερη σημασία σε ομάδες μη προνομιούχων ανθρώπων, ατόμων. Συχνά οι ομάδες που θα υποφελούνταν περισσότερο μένουν σε αυτό το 5% αντί να αυξάνεται η συμμετοχή καθεαυτήν, να αυξάνουμε τη συμμετοχή καθεαυτήν, οι χώρε μέλη θα έπρεπε να διευρύνουν τη συμμετοχή ώστε να περιλάβει και ομάδε που είναι δυσπρόσιτε, με ειδικέ ομάδε στόχου. Παιδιών, για παράδειγμα, σε περιοχέ τη Υπέθρου. <clears throat> Βλέπουμε αρκετέ ενδείξει στη μελέτη αλλά και στη βιβλιογραφία για μια ανάγκη υιοθέτηση μιας τάσης ε, ενοποίησης των δομών οι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων για την πολιτική για τα πιο νέα παιδιά, για τα πιο νεαρά παιδιά, θα πρέπει να είναι σε επαφή με τους αρμόδιους για την εκπαίδευση συνολικά, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για την ανάπτυξη των παιδιών. Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο θα υποστηρίζει τους παρόχους των υπηρεσιών για να βελτιώνουν διαρκώς τις υπηρεσίες τους. Διότι μέχρι τώρα υπάρχουν προδιαγραφές, ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας. Αυτό δεν αρκεί. Μια κρίσιμη απέτηση τώρα είναι και το προσωπικό που πρέπει να, είναι, να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και εξοπλισμό. Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις στη μελέτη που καθιστούν απαραίτητο να απαιτούνται κάποιες, κάποια ελάχιστα προσόντα για παράδειγμα από την ε, εκπαίδευση για ένα μείγμα ε, ανώτερη εκπαίδευσης και επαγγελματική εκπαίδευσης. Όσο πιο εκπαιδευμένο το προσωπικό, τόσο μεγαλύτερη ποιότητα, τόσο καλύτερη ποιότητα προσφέρει. Για να υποστηριχθούν αυτές οι εξελίξει πολιτικής, είναι σημαντικό οι ε, χώρε μέλη να εμένουν σε απαιτήσει του, αλλά και να προβλέπουν την απαραίτητη χρηματοδότηση. Δεν αρκεί δηλαδή να αυξάνουν τι απαιτήσει προσόντων του προσωπικού χωρί να προσφέρουν σχετική χρηματοδότηση. Πρέπει λοιπόν να, να υλοποιήσουν τι δεσμεύσει του και τελικά δηλαδή να ε, κάνουν έργο τα λόγια του. Είναι σημαντικό επίση να ληφθεί υπόψη και να μην υποτιμηθεί η επίπτωση της δημοσιονομικής κρίσης. Οι περικοπές των προϋπολογισμών για την ε, φροντίδα των ε, μικρών στερεί τα απαραίτητα από τις ομάδες που τα έχουν περισσότερο ανάγκη. Θα πρέπει λοιπόν οι να δράσουν αναλόγως. Τέλος, θα ήθελα να θυμίσω τα λόγια του James Hackman, νομπελίστα οικονομολόγου, που λέει ότι κάθε ευρώ που ξοδεύει κανείς για τη φροντίδα της νεαρότατης ηλικίας είναι, αποδίδει πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη επένδυση στην εκπαίδευση και ιδίω για μη προνομίωσες ομάδες. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η φροντίδα της νεαρής ηλικία σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Δηλαδή. Ευχαριστώ κύριε Λίντεμπουργκ και τώρα έχουμε βέβαια πολλούς που ενδιαφέρονται να λάβουν το λόγο. Κύριε Χάνιμπαλ πρώτη. Ναι, ευχαριστώ. Πραγματικά ευχαριστώ. Ήταν μια έκθεση που πήγε πραγματικά σε βάθος και ευχαριστώ για όλη τη δουλειά που κάνατε. Είναι ενθαρρυντικό, γιατί άλλωστε και εγώ στην έκθεσή μου στα ίδια συμπεράσματα καταλήγω, ενθαρρυντικό ότι υπάρχει συμφωνία για την κρίση της κατάστασης σε ολόκληρη την Ένωση. Μου άρεσε που μιλήσατε για την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, διότι χρειάζεται κάτι να κάνουμε. Συχνά λαμβάνουμε εκθέσεις που είναι πολύ ενδιαφέρουσες και καταστρώνουν πολύ ωραία τα γεγονότα και τις ιδέες, αλλά δεν καταλήγουν πουθενά. Νομίζω το θέμα είναι τόσο σημαντικό που είναι αδύνατο να αγνοηθεί. Εσείς νομίζω μας υποδεικνύετε έναν τρόπο που μπορούμε να υιοθετήσουμε απέναντι στις χώρες μέλη, γιατί βέβαια είναι ένα θέμα δική τους αρμοδιότητα είναι και όχι δική μας. Άρα χρειάζεται να γίνει μέσα από τη μέθοδο ανοιχτού συντονισμού και χαίρομαι που δίνεται ιδιαίτερο βάρος σε αυτό. Και νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να προχωρήσουμε. Πιθανώς στο προσεχές μέλλον να μην μπορέσουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. έτσι ώστε να προσεγγίσουν τα συστήματα που εφαρμόζουν διάφορε χώρε μέλη. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να κάνουμε αυτό. Όσο υπάρχει κάποια συνεκτικότητα στην ποιότητα και οι χώρε μέλη έχουν όλε ένα στόχο βελτίωση, δεν έχει ίσω σημασία το ότι οι χώρε μέλη προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο το θέμα η καθεμιά. Χαίρομαι λοιπόν για την έκθεση αυτή. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε τώρα στην Επιτροπή Πολιτισμού είναι να παραμείνουμε στο παιχνίδι, να ενθαρρύνουμε την επικοινωνία, να εξετάζουμε την κατάσταση της χώρας μέλη, καθώς προχωρούμε, και με λίγα λόγια σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Μπόρις. Ευχαριστώ, αγαπητή Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ε, μελέτη Αυτό που λείπει στις χώρες μέλη είναι συγκριτικές μελέτες. Εγώ έχω τρία παιδιά. Και με τα παιδιά μου ορισμένα, μάλλον ε, ε, έχω δηλαδή περάσει ε, ήδη αυτή την πρώτη ηλικία, αλλά είναι και ένα που είναι ακόμα σε αυτή την ηλικία και είναι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό το θέμα αυτό. Και για την Πολωνία βρίσκω ότι η πρόσβαση σε αυτές τις ε, φροντίδες, σε αυτές τις υπηρεσίες είναι, είναι, ε, είναι ε, καλή. Με την στήριξη των αρμόδιων ταμείων μπορούν να δημιουργηθούν και χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς και κυρίως σε τόπους, μικρές πόλεις και γενικά στην Ήπεθρο όπου δεν υπήρχαν τέτοιες υπηρεσίες. Και το θέμα τώρα της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Καθώς επίσης τις επιρροή που έχουν τα παιδιά στην σταδιοδρομία των γυναικών είναι σημαντικά. Σε πολλές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης πρέπει να δημιουργηθούν οι υπηρεσίες αυτές υπερομάδων που δεν είχαν την δυνατότητα αυτή στο παρελθόν. Εκεί η ποιότητα είναι πολύ σημαντική. Μιλούμε για παιδιά ηλικία 3 6 ετών, τουλάχιστον στην Πολωνία. Ακόμα τα παιδιά δεν είναι υποχρεωμένα να πάνε στο σχολείο. Οι γονεί συχνά προτιμούν να τα αναθέσουν στη φροντίδα των παππούδων ή ένας από τους γονιούς μένει στο σπίτι αλλά πρέπει να επιμείνουμε ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα. Έχω δει ε, νηπιαγωγεία που εφαρμόζουν τις μεθόδους Βάλντορφ, άλλα Μοντεσόρι, που κάνουν τα παιδιά πιο υπεύθυνα για τους εαυτούς τους. Υπάρχουν και νηπιαγωγεία όπου τα παιδιά τους μιλούν σε τρεις γλώσσες, για παράδειγμα σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας μου. Υπάρχουν ε, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, όπου διδάσκονται παιδιά, δηλαδή ε, Πολωνάκια και Γερμανάκια ταυτόχρονα. Όμως δεν υπάρχει σύστημα προώθησης της ποιότητας, της προώθησης των βέλτιστων πρακτικών. Δεν υπάρχει μηχανισμός σύγκρισης που να επιτρέπει να συγκρίνει κανείς πώς δαπανώνται τα κονδύλια αυτά. Ωστόσο αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να πείσουμε και τους, γεγον... και, τους γονείς ότι δεν είναι μόνο η διαθεσιμότητα ε, θέσεων στους παιδικούς σταθμούς, αλλά και η ποιότητα. Είναι δύσκολο να προσεγγίσει κανείς τις χώρες μέλη, διότι σε πολλές χώρες, όπως για παράδειγμα στην Πολωνία, δεν είναι το κράτος αρμόδιο, αλλά οι κοινότητες. Άρα συνομιλητές μας θα έπρεπε, δεν θα είναι μοιραία τα κράτη, αλλά οι χιλιάδες των κοινοτήτων Νομίζω ότι ε, χρειάζεται να ασκηθεί ακόμα πολύ μεγαλύτερη πίεση για να βελτιωθεί η ποιότητα. Μαρή Τερέζ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ την Επιτροπή ότι αφιέρωσε τόσο χρόνο σε ένα από τα θέματα που δεν μας απασχολούσαν ιδιαίτερα, δεν ήταν στις προτεραιότητές μας εδώ και λίγο καιρό, που τώρα αποτελεί κύριο μέλημα των κρατών μελών. Γνωρίζουμε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς μία ανταγωνιστική οικονομία μέσα στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 και είναι σίγουρο ότι η έρευνα και η καινοτομία ε, είναι ε, μίζονες προτεραιότητες ε, διότι αποτελούν πόλο έλξης και αριστείας. Πρόκειται για έναν τομέα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για μια δελεαστική οικονομία, δηλαδή την έρευνα όπου γίνεται λόγος για εκπαίδευση και προσχολική ηλικία Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η υποδοχή των ε, μικρών παιδιών. Επιμείνατε στο θέμα της ποιότητας. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να φτάσουμε σε έναν ευρωπαϊκό ορισμό ε, του, του θέματος αυτού. Εν πάση περιπτώσει η μελέτη σας μας επιτρέπει να φτάσουμε σε μία ιχνηλάτηση ως προς την προσχολική ηλικία και βεβαίως ε, πρόκειται για θέμα εθνικής προτεραιότητας. Πώς μπορούμε να μιλήσουμε για εκπαίδευση ποιότητας, μπορούμε να μιλήσουμε για ελάχιστες προδιαγραφές, πώς ε, τις ορίζουμε όπως ισχύει με τις ε, ζωντανές γλώσσες. Δεν έχουμε επαρκή στοιχεία γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς η προσχολική ηλικία μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν μπορεί να μετρηθεί επαρκώς, είναι όμως ένας τομέας στον οποίο μπορούμε να παρέμβουμε ιδιαίτερα με αξιολογήσεις που επιτρέπουν στη συνέχεια να κρίνουμε πώς ε, ε, αντιμετωπίζεται η προσχολική ηλικία και πώς μπορεί αυτό να αποτελέσει ε, κάτι το θετικό για το μέλλον. Ως προς τη Γαλλία έχουμε ένα πολύ καλά οργανωμένο σύστημα υποδοχής για την προσχολική ηλικία. Υπάρχουν βρεφονιπιακοί σταθμή όπου υπάρχει συντονισμός σε εθνικό επίπεδο, καθώς και νηπιακή σταθμή, καθώς και στοιχεία ε, συνοδευτικά, δεν ξέρω ποιο προϋπήρξε ε, η κότα ή το αυγό. Θα πρέπει να δούμε και τον ε, δίκτυ εθνισιμότητας, ο οποίος όμως είναι ο πιο υψηλός στην ε, Ευρώπη. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει μια διτή προσέγγιση, όπως είπατε, καταρχήν ε, η εκπαιδευτική προσέγγιση αλλά και η κοινωνική, διότι η προσχολική ηλικία αφορά ένα επίπεδο, ε, επίπεδο αντιμετώπισης και της επισφάλειας που υπάρχει σε επίπεδο κοινωνίας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς ε, υπάρχει και αν υπάρχει καλή κατανομή σε περιφερειακό επίπεδο, κάτι το οποίο δεν ισχύει και θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά κάτω από τριών ετών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την μελέτη και είμαι σίγουρη ότι αυτά τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά για μια μελλοντική συνεργασία. Δεν υπάρχουν ε, ε, μαγικές λύσεις, αλλά θα πρέπει να προβούμε σε ανταλλαγή ε, πρακτικών και ένας προγραμματισμός για τα κράτη που θέλουν να θέσουν σε εφαρμογή συστήματα που δεν υπάρχουν. Μιλήσατε για, για, για πολιτική συμμετοχή. Η απάντηση είναι σαφής. Το πρώτο που μας απασχολεί είναι η χρηματοδότηση. Καμία πολιτική δεν μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή χωρίς χρηματοδότηση. Ως προς την ε, κατάρτιση, εάν δεν υπάρχει ε, επαρκής ποιότητα, τότε θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο επίπεδο της κατάρτισης και να προωθήσουμε μία ε, πολιτική θέληση σε επίπεδο κρατών μελών. Η χρηματοδότηση έχει μεγάλη σημασία και τα περιφερειακά ταμεία και η πολιτική θέληση για να ε, υποβάλουμε πολιτικές σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστούμε τα Μαρή Τερέζ και, το, και τώρα η Σίλβια. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα μελέτη. Όπως είπε και η συνάδελφος η Μαρία Χάνιμπαλ και όπως είπε και ο ερευνητής μας, θα πρέπει να προχωρήσουμε λίγο πιο μακριά. Γιατί εδώ έχουμε κατευθυντήριες γραμμές και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να γίνουν γενικότερες συστάσεις. Θα ήθελα να μιλήσουμε και για την ποιότητα είναι γεγονός ότι μας ενδιαφέρουν ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα συστατικά στοιχεία αυτής της ποιότητας. Δηλαδή, να μιλήσουμε για μια ενιαία υπηρεσία και συλλογική εργασία από πλευράς εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών αρχών. Ένα άλλο σημαντικό είναι η ενημέρωση του προσωπικού. Δηλαδή να υπάρχει ένα ε, γενικό πρότυπο προδιαγραφών. Επίσης μιλάμε για προσωπικό, επαγγελματικό προσωπικό και ε, παιδιά. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει μια σωστή ε, ποσοστή αναλογία, δηλαδή κατά πόσο αριθμητικά επαρκεί αυτό το προσωπικό. Μας ενδιαφέρει και το θέμα των παιδιών με ε, αναπηρίες γιατί θα ήθελα να ξέρω ε, πώς αντιμετωπίζεται από άλλες χώρες. Ως προς το θέμα της ολοκλήρωσης δεν κατάλαβα την πρότασή μας. Είπατε ότι οι υπηρεσίες για τα μικρά παιδιά, δηλαδή η προσχολική ηλικία, θα πρέπει να αποτελεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία. Μιλάτε για 0 έως 6 χρόνια. Αυτή είναι η παιδαγωγική αρχή. Νομίζω ότι θα πρέπει η ενσωμάτωση να αφορά και, και το δημοτικό. Δηλαδή μιλάμε για προσχολική ηλικία και ε, δημοτικό. Να υπάρχει σωστή μετάβαση γιατί τα παιδιά δεν είναι πακέτα που τα στέλνουμε στο σχολείο. Θα πρέπει η προσχολική εκπαίδευση να προετοιμάζει προς, τον, προς την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μιλήσατε για το ηλικιακό φάσμα 0-6 χρόνια. Θα πρέπει να δούμε τι ευκαιρίες δημιουργούνται. Γιατί και στη χώρα μου βλέπουμε ότι τα παιδιά 2-3 ετών ενσωματώνονται καλύτερα. Ε, πολλές μικρές χώρες όμως δεν δημιουργούν επαρκείς βρεφονιπιακούς σταθμούς. Ε, στα 2-3 χρόνια υπάρχουν υποδομές υποδοχής, αλλά υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τα τρία στα έξι χρόνια. Θα ήθελα μία διασάφηση εδώ και να δούμε και τις επιπτώσεις της κρίσης. Είδαμε σε πολλές χώρες, όπως και στη δική μου, μία συρρήκνωση των υποδομών. Θα ήθελα να μας πείτε πώς η κατάσταση. Τα παιδιά επίσης που ε, εισάγονται πολύ νωρίς, που μπαίνουν πολύ νωρίς στον βρεφονιπιακό σταθμό δεν, έχουν καλά, δεν δείχνουν καλά αποτελέσματα. Δηλαδή όταν για λόγους αναγκαιότητας τα παιδιά τα πάμε σε ένα βρεφονιπιακό ή βρεφικό σταθμό στους πέντε μήνες μετά δεν τα καταφέρνουν και τόσο καλά. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε και μία παιδαγωγική προβολή της ε, κοινωνικοποίησης των παιδιών. Δηλαδή, τι γίνεται με τα παιδιά τριών έως έξι ετών, τα οποία δεν είχαν εισαχθεί σε έναν βρεφικό σταθμό από τους πέντε μήνες. Ε, ευχαριστώ. Να προσθέσω κάτι ακόμη, λέει η πρόεδρος κυρία Πακ. Ξαφνιάστηκα όταν είδα που βρίσκεται η Φιλανδία στην υπόθεση αυτή που έχει τον μικρότερο αριθμό, τον μικρότερο ποσοστό παιδιών ενώ η Πίζα λέει ότι είναι η καλύτερη στα αποτελέσματα των εξετάσεων. Διάβασα όμως ότι στη Φιλανδία είναι βέβαιος η διαδεδομένη άποψη ότι το καλύτερο είναι να μην να ευγίνονται με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή το κράτο πληρώνει και δασκάλου και όλα. Και αυτά ίσω να τα διάβασε και η Τσέσου όταν αποφάσισε τα σχετικά με την κατάργηση του επιδόματο φροντίδα. Τώρα, όπω είπε και του, η εκμάθηση γλώσσα όταν τα παιδιά είναι πάρα πολύ μικρά. Είναι πολύ σημαντικό. Το θέσατε το θέμα αυτό. Δεν το βλέπω στο κείμενο ή σας φάνηκε αμελητή αποσότητα. Διότι όταν, για παράδειγμα, κάποιοι κατοικούν σε παραμεθόριες περιοχές, όπως στο Γκέρλιτς ο φίλος μας από την Πολωνία ή εγώ που είμαι στο Σάρλαντ, στα γαλλογερμανικά σύνορα. Είναι πολύ κρίμα να μην μάθει κανείς τη γλώσσα του γείτονα και μάλιστα με τρόπο σαν παιχνίδι ας πούμε και όσο γίνεται νωρίτερα. Επομένως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει σε παιδικούς σταθμούς με διαφόρους τρόπους. Δεν μιλούμε για δογματική ε, ε, διαπαιδαγώγηση, αλλά μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι μιλούν τη γλώσσα αυτή ως μητρική τους και την μεταφέρουν στο παιδί. Αναρωτιέμαι λοιπόν εάν κάπου το έχετε λάβει υπόψη σα αυτό στη μελέτη σα ή όχι. Άλλε ερωτήσεις? Εσεί. Ευχαριστώ για την ε, παρουσίαση της μελέτης σας. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Θα ήθελα να μας πείτε περισσότερα για την συμμετοχή ευάλωτων μη προνομιούχων ομάδων στην ε, εκπαίδευση πολύ νεαρή ηλικία. Στη Σλοβακία έχουμε σημαντικά προβλήματα για να πετύχουμε να μπουν στην προσχολική εκπαίδευση τα παιδιά των Ρώμα. Δεύτερο, γιατί επιλέξατε τις έξι αυτές συγκεκριμένες χώρες για την μελέτη, για τις case studies. Είδαμε έκπληξη ότι μόναχα μία ανατολική χώρα, η Ρουμανία, ε, περιλαμβάνεται μεταξύ αυτών. Ωστόσο, οι ανατολικές χώρες της Ευρώπης έχουν κάποια προβλήματα που ε, προκύπτουν από την μετάβαση από το κομμουνιστικό καθεστώς σε άλλα καθεστώτα. Γιατί έκλεισαν τότε πολλοί παιδικοί σταθμοί και τώρα μας λείπουν. Νομίζω ότι έχει νόημα να συγκριθεί η κατάσταση στην Ανατολική Ευρώπη με αυτή της Δυτικής Ευρώπης. Άλλωστε συμφωνώ με την Τόρις σε ό,τι αφορά την γλωσσική παιδεία. Στην Σλοβακία τα περισσότερα σχολεία μαθαίνουν στα παιδιά τα αγγλικά σαν παιχνίδι. Εσείς μιλήσατε και για ποσοτικά και για ποιοτικά στοιχεία και τονίσατε ιδιαίτερα την ανάγκη της ποιότητας. Ωστόσο εμένα μου φαίνεται ότι και η ποσότητα παίζει ρόλο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν μέρη όπου είναι μεγάλο πρόβλημα να βρεθούν παιδικοί σταθμοί ή τέλος πάντων κέντρα προσχολικής εκπαίδευσης. Και υπάρχει και διαφορά ανάμεσα σε αυτές που χρηματοδοτούνται από το κράτος και αυτές που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές. Πρέπει ε, στην προσπάθεια αυτή για την προσχολική εκπαίδευση να συμμετάσχουν περισσότερο και το διδακτικό προσωπικό. Επίσης το συνολικότερο ύφος της μελέτης ή μάλλον επιτρέψτε μου να διορθώσω λίγο αυτό που θέλω να πω. Μιλώ περισσότερο για τη γλώσσα που νομίζω ότι είναι πρόβλημα να βρει κανείς μια μελέτη σε γλώσσα άλλη εκτός από τις τρεις τέσσερις μεγάλες γλώσσες όπως λέγονται. Εγώ μπορώ να διαβάσω βέβαια ε, κάποιες μελέτες στα αγγλικά, αλλά τουλάχιστον κάποιες μελέτες θα έπρεπε να εκδοθούν και σε άλλες γλώσσες, ανατολικοευρωπαϊκές ας πούμε. Πάντως σας ευχαριστώ. Είχε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον η μελέτη. Να προσθέσω κάτι ακόμη. Γιατί χρησιμοποίησατε δεδομένα του 2010 και του 2000 Ίσως θελήσατε να λάβετε ως βάση της σύγκρισης την δεκαετία. Δεν θα έπρεπε να εξετάσετε και τα πιο πρόσφατα έτη, για παράδειγμα το 2012 σε σύγκριση με το 2002. Και εγώ θα ήθελα να σταθώ στην διδαχή των γλωσσών αυτό το θέμα μας απασχολεί σε τακτά χρονικά διαστήματα υπό μία άλλη προοπτική, διότι εμείς είμαστε τραγικοί στην διδασκαλία των γλωσσών. Θεωρούμε ότι δεν χρειάζονται Νομίζω ότι τα παιδιά χάνουν από την μη διδασκαλία, την έλλειψη διδασκαλίας ε, ξένων γλωσσών. Θα πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσει αυτό το θέμα, να υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή φιλοδοξία, δηλαδή τα παιδιά να μιλάνε δύο άλλες γλώσσες εκτός από τη μητρική. Αν και δεν συμβαίνει ε, στη Βρετανία, στη Μεγάλη Βρετανία κάτι τέτοιο, ούτε προβλέπεται από τα μαθήματα. Υπάρχουν πολλές πτυχές ε, στη διδασκαλία και αν θέλουμε αυτή την έκθεση να τη δούμε ως μία ε, μεθοδολογική προσέγγιση και ε, προσέγγιση συντονισμού θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε εμείς τα τρία μέλη της Επιτροπής, κατά πόσο μπορεί δηλαδή να εισαχθεί ε, στο πρόγραμμά μας όπως έχει οριστεί. Υπάρχει κάποιος από την Επιτροπή που θα ήθελε να παρέμβει, όχι. Για την μετάφραση βεβαίως κύριε Λίντεμπομ δεν είστε εσείς ε, υπεύθυνο ε, οφείλεται στον προπολογισμό μας αυτό. Άλλε ερωτήσει. Όμως μπορείτε να απαντήσετε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ακούστηκαν πολλά, πολλές ενδιαφέρουσες απόψεις. Θα ξεκινήσω με τις παρατηρήσεις σχετικά με την ενοποίηση των δομών. Αυτό που προσπαθήσαμε να δείξουμε και να προωθήσουμε είναι πώς αυτές οι διαφορετικές ε, μονάδες ε, προσχολικής εκπαίδευσης μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα. Υπόθηκε ότι ε, ενδεχομένω δημιουργούμε ένα καινούριο όριο στην ηλικιακή ομάδα 0 έως 6. Το επιλέξαμε αυτό αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ήταν σκοπός μας να δημιουργήσουμε ένα νέο ηλικιακό φράγμα. Η μελέτη στην ουσία επιβεβαιώνει ότι τα, οι φορείς αυτοί θα πρέπει να συνεργάζονται με δομές προσχολικής εκπαίδευσης, ε, παροχής υγείας. Το μήνυμα λοιπόν το βασικό μήνυμα είναι ότι η συνεργασία μεταξύ αυτών των ε, οργάνων, μεταξύ αυτών των φορέων είναι, είναι εξαιρετικά σημαντική για την ποιότητα στην προσχολική εκπαίδευση. Το ερώτημα για το πότε πρέπει να πάει ένα παιδί στον παιδικό σταθμό. Στην μελέτη δεν προσπαθήσαμε να ε, κάνουμε κάποια υπόδειξη, ε, είναι επιλογή των γονέων. Σε κατά κύριο λόγο ε, εξαρτάται και από τον πολιτισμό, από την κουλτούρα ε, που κυριαρχεί σε κάθε χώρα. Αναφερθήκατε και στην Φιλανδία όπου ε, η επιλογή της, του, του να μην πάνε τα παιδιά στο σχολείο θεωρείται η καλύτερη επιλογή. Παρ' όλα αυτά οι γονείς είναι εκείνοι που κάνουν την επιλογή. Προσπαθήσαμε λοιπόν να μην εκφράσουμε κάποια πολύ αυστηρή θέση όσον αφορά ε, το ζήτημα αυτό. Θα πρέπει να αποφασίζεται δηλαδή στο ε, χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Όσον αφορά το προσωπικό, για την ε, ε, διαρκή εξέλιξη των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού, πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε δηλαδή την συνεχή βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό. Στην μελέτη συμπεριλάβαμε, βεβαίως Τώρα στην παρουσίαση ήμουν πολύ σύντομο και δεν μπόρεσα να καλύψω όλα τα ζητήματα που εξετάσαμε. Πάντως εξετάσαμε σε ποιο βαθμό τα κράτη-μέλη ε, έχουν θεσπίσει τέτοιου κανόνες για την ε, υποχρεωτική ε, επαγγελματική, διαρκή επαγγελματική μετεκπαίδευση για το προσωπικό. Κάποια κράτη-μέλη έχουν ένα πιο προαιρετικό σύστημα, να το πω έτσι, για τα μέλη του προσωπικού. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια συνολική εικόνα, μια επισκόπηση του τι συμβαίνει. Τώρα, για ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που ακούστηκε. Οι γλωσσικές δεξιότητες που αναφέρθηκαν από πολλούς. Δεν εστιάσαμε στο ζήτημα αυτό στην έκθεσή μας, διότι και οι χώρες που επιλέξαμε, για παράδειγμα στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, στη Γερμανία, ε, ε, υπάρχουν ενδεχομένως κάποια δίγλωσσα σχολεία. Στην Φιλανδία πάντως μιλήσαμε με ε, ένα ίδρυμα που προσφέρει αγγλική εκπαίδευση και ε, μας παρέσχει μια πολύ ενδιαφέρουσα οπτική. Ωστόσο, έχουμε και, κάναμε και μια άλλη παρατήρηση στην ε, μελέτη, ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ε, εστίαση στην εκπαίδευση. Και ε, είπαν και πολλοί εδώ ότι είναι σημαντικό να μαθαίνονται, να διδάσκονται γλώσσες με έναν, σαν παιχνίδι και να... Ε, φυσικά η συμπερίληψη της δασκαλίας ξενογλωσσών γλωσσών μπορεί να έχει πλεονεκτήματα αλλά μπορεί να έχει και μειονεκτήματα διότι μπορεί να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα τάξης σχολικής και ε, ε, να υπενθυμίσω ότι ενδεχομένως το να μην πάει το παιδί στο σχολείο είναι ίσως η καλύτερη επιλογή για τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού. Τώρα, για τις ξένες γλώσσες και τις γλωσσικές αξιότητες συμπεριλάβαμε υπόψη μας και την ε, φιλανδική εμπειρία, τη φιλανδική πρακτική και ναι, πάντως είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα αυτό που θέσατε. Τέθηκε ένα ερώτημα σχετικά με το ποια κριτήρια χρησιμοποιήσαμε για την επιλογή των χωρών που μία ανατολικοευρωπαϊκή χώρα. Συμφωνώ απολύτως ότι υπάρχει βεβαίως μια ανατολικη ευρωπαικη χωρα συμφωνω απολυτως οτι μεταξύ των παλαιών και των νέων κρατών μελών. Πάντως στην ε, μελέτη προσπαθήσαμε να ενσωματώσουμε διάφορες ε, ομάδες ε, και διάφορες κουλτούρες εκπαίδευσης. Οι χώρες που έχουν ε, κομμουνιστικό παρελθόν και προσπαθούν να αναδιαρθρώσουν τις ε, δομές προσχολικής ε, εκπαίδευσης ανέδειξαν, είναι ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Εξετάσαμε και την κουλτούρα, την εκπαιδευτική κουλτούρα που ε, κρύβεται πίσω από την ανάπτυξη συγκεκριμένων πολιτικών. Ε, προσπαθήσαμε δηλαδή ε, να καλύψουμε και γεωγραφικά την Ευρώπη για να αντικατοπτριστεί και με κάποιον τρόπο και ε, να αντικατοπτριστούν και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις χώρες. Αυτά ήταν εν πολλής τα κριτήρια επιλογής των χωρών. Φυσικά θα, και, θα μπορούσαμε και θα ήταν και πολύ ενδιαφέρον να, να είχαμε επιλέξει και άλλες πολλές χώρες. Αλλά αυτή ήταν εν τέλει η επιλογή χωρών που κάναμε Επίσης ακούστηκε ότι εκτός από την ε, έμφαση στην ποιότητα η ποσότητα είναι σε κάθε περίπτωση σημαντικά. Βεβαίως συμφωνούμε. Απλά αυτό που τονίζουμε στην έκθεσή μας είναι ότι η ποσότητα από μόνη της δεν είναι κάτι που από μόνο του αξίζει να υπάρχει ως στόχος. Αλλά βεβαίως η πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης είναι σημαντικό ζήτημα. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση να συγκριθούν ε, οι φορείς που χρηματοδοτούνται και εκείνοι που δεν χρηματοδοτούνται από το κράτος. Την είχαμε εξετάσει και εμείς αυτή την ιδέα. Αλλά ε, ο κύριος στόχος μας, ε, η κύρια εστίασή μας στην μελέτη αυτή ήταν οι κρατικά χρηματοδοτούμενοι φορείς. Αλλά πάντως συμφωνώ θα ήταν πράγματι μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή για μια ενδεχόμενη μελλοντική μελέτη και με πολύ ενδιαφέρον θα περιμέναμε τα αποτελέσματα. Τώρα, για, το, για την περίοδο 2000-2010 ε, που επιλέξαμε, ε, πήραμε τα πιο ε, πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα από τη Eurostat που αφορούσαν το 2010 και όπως τονίστηκε ναι, πράγματι προσπαθήσαμε να, να εξετάσουμε μια ε, ε, δεκαετία για να καλύψουμε και την περίοδο πριν την ε, θέσπιση συγκεκριμένων ε, στόχων. Η θέσπιση των στόχων έγινε το 2002, υπενθυμίζω. Γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε αυτό το χρονικό διάστημα. Και ένα τελευταίο σημείο τέθηκε νωρίτερα είναι η σχέση μεταξύ του προσωπικού και των παιδιών. Ένα επίσης πολύ σημαντικό ζήτημα που εξετάζουμε και στην έκθεσή μας. Προσπαθούμε να δείξουμε πόσοι οι καθηγητές, πώς οι δάσκαλοι υπάρχουν ε, στο προσωπικό. Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα στοιχεία από τα κράτη-μέλη. Ε, πάντως η μέθοδος μέτρησης σε κάθε κράτος μέλος διαφέρει και θα ήταν καλό ε, αν μπορούσαμε τουλάχιστον να συγκρίνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτές τις μεθόδους μέτρησης να δούμε δηλαδή ποια είναι η αναλογία προσωπικού και παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δυστυχώ η μελέτη όμως δεν αφορούσε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά μόνο τα έξι αυτά που επιλέξαμε. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Ήταν πολύ χρήσιμη η συζήτησή μας. Ευχαριστώ που συμμετείχατε, αγαπητοί συνάδελφοι. Να προχωρήσουμε στο σημείο 9. Νέε τεχνολογίε και ανοιχτή εκπαιδευτική πόρη. Ήβαν, σα παρακαλώ, κλείστε το τηλέφωνο σα. Είστε ο εισηγητή. Λοιπόν, τι θέλετε να μα πείτε. Καταρχήν, Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να ε, μιλήσω για αυτή την έκθεση διότι είναι ένα θέμα ύψης της σημασίας. Η οικονομική κρίση, τα διεθνή δεδομένα, ο ανταγωνισμός των μεγάλων οικονομικών μπλοκ Ασίας, Ευρώπης, Αμερικής, Νότιος Αμερικής ε, μας απασχολούν ιδιαίτερα. Επίσης, η ενδογενής μας οικονομική κρίση, η ανεργία των νέων, η ενή αγορά η αγορά απασχόλησης, όλα αυτά αποτελούν μία απτή πραγματικότητα. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε την γενεά των εργοδοτών και των νέων στα πανεπιστήμια. Το θέμα λοιπόν των νέων τεχνολογιών και των εκπαιδευτικών πόρων αποτελεί μια απτή πραγματικότητα και μας ενδιαφέρει η καλύτερη δυνατή χρήση αυτών για την επίλυση βασικών ζητημάτων. Το 50 με το 80% των ε, μαθητών ε, και ε, εκπαιδευτών δεν χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα. Επίσης, οι δάσκαλοι και καθηγητές του, ε, της πρωτογενούς και δευτερογενούς εκπαίδευσης δεν χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους. Η εκπαίδευση βασίζεται στη, στους παραδοσιακούς τρόπους ε, μελέτης και διδαχής. Δηλαδή, οι μαθητές δεν χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες, δεν χρησιμοποιούν ε, τα, ε, τις οδηγίες χρήσης δεν χρησιμοποιούν επαρκώς το διαδίκτυο. Δεν χρησιμοποιούν τις επιγραμμικές υπηρεσίες, ενώ θα έπρεπε να χρησιμοποιείται αυτή η πληθώρα πληροφοριών και στην Αμερική και στην Ασία και στην Ευρώπη. Τα ε, περισσότερα δελτία και οδηγίες χρήσης υπάρχουν στα αγγλικά. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η εργατική δύναμη να είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένη ε, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κοινωνίας μας. Μιλάμε και για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα 2020, μια οικονομία που βασίζεται στη μελέτη και στη γνώση. Αντιμετωπίζουμε ε, τρεις προκλήσεις. Καταρχήν ότι δεν υπάρχει καινοτομία στον εκπαιδευτικό τομέα. Η δεύτερη πρόκληση είναι η ανεπαρκής χρήση των εκπαιδευτικών πόρων, των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων και τρίτον η έλλειψη υποδομών έτσι ώστε το διαδίκτυο να μπορέσει να μπορεί να χρησιμοποιείται από όλους τους μαθητές. Και εδώ αναφέρομαι στο διαδίκτυο και στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας. Οι προτάσεις της Επιτροπής είναι τρεις. Η αναγνώριση της χρήσης διαδικτύου και επιγραμμικών υπηρεσιών και επίσης η ψηφιακή κοινωνία, ε, προσβασιμότητα στο εκπαιδευτικό ε, υλικό και βελτίωση των ευρυζωνικών υπηρεσιών του διαδικτύου σε επίπεδο ε, μαθητείας. και στις τάξεις του σχολείου. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, διότι η προσβασιμότητα θα έπρεπε να εξασφαλιστεί, να είναι εξασφαλισμένη, ιδιαίτερα ως προς τις σύγχρονες τεχνολογίες της επικοινωνίας για τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και την ομοιογενοποίηση της ποιότητας και του υλικού των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων. Όλα αυτά θα μπορέσουμε να τα αποτιμήσουμε στο μέλλον. Πιστεύω επίσης ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ουραγός έμπρακτα των ΗΠΑ ή της Ασίας, εκεί όπου γίνονται επενδύσεις στη σύγχρονη τεχνολογία επικοινωνίας. Και επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να διενεργηθεί μία μελέτη γιατί δεν ξέρω αν προϋπάρχει, για να δούμε ποια είναι η σχέση μεταξύ παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας και σύγχρονων. Γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες, αλλά ίσως υπάρχουν μελέτες ε, τις οποίες θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και δεν χρειάζεται να απαρνηθούμε όλες τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Απλώς πρέπει να φτάσουμε σε μία σωστή ισορροπία μεταξύ των ε, δύο. Να δούμε μέχρι πού θα φτάσουμε με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών και τι επιθυμούν οι νέοι με τη λήξη των σπουδών όταν μιλάμε για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Επίσης, ποιες είναι οι απαιτήσει της αγοράς εργασίας και τι ανάγκες θα υπάρξουν στο εγγύς μέλλον. Tą prezentację, ona, ona tak naprawdę dotyka Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θέσατε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων σε σχέση με τις μεγάλες προκλήσεις στο τομέα διδασκαλίας στα σχολεία, διότι μας ενδιαφέρουν οι ανάγκες των μαθητών αλλά και του διδακτικού προσωπικού. Μιλάμε για μια νέα γενιά, τη γενιά της πληροφορίας και της πληροφορικής Πολλές φορές χρειαζόμαστε πληροφορίες από το διαδίκτυο, χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα, αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε επαρκώς. Και αυτό αφορά και το διδακτικό προσωπικό, μέσα στα πλαίσια της επικοινωνίας, της επικοινωνίας που εξασφαλίζει το διαδίκτυο. Πολλές φορές Υπάρχουν πληροφορίες στο διαδίκτυο και πολλές φορές λένε οι καθηγητές μεταξύ τους «Α, κοίταξε, αδές αυτό το σημείο, διότι όπως βρήκα στο διαδίκτυο ε, υπάρχει αυτή η εξέλιξη στον τομέα ή το δίδαξες λάθος». Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μία σωστή πρόσμιξη μεταξύ του παραδοσιακού συστήματος διδασκαλίας και των ε, νέων τεχνολογιών που μπορούν να βοηθήσουν ιδιαίτερα. Δεν μιλάμε μόνο για τα προσόντα που προϋπάρχουν, αλλά μας ενδιαφέρει και η ε, σωστή χρήση του διαδικτύου, διότι μιλάμε για μία ε, ζούγκλα πληροφοριών, μία πολυμηνυματική κοινωνία και θα πρέπει να γίνει σωστή χρήση του διαδικτύου, δηλαδή να λάβουμε υπόψη και την αρχή της επιλεξιμότητας. Πολλές φορές έχουμε εξαιρετικούς ε, καθηγητές και στον τομέα του e-learning. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει διάδραση, η χρήση και του πίνακα και του διαδικτύου. Αυτό ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα και να γίνει σωστή χρήση και των ε, χρηματικών πόρων και αυτό για τη νέα γενιά. Δηλαδή τα παιδιά μου 6 και 7 ετών ήδη καν παρουσιάσει σε PowerPoint. Δηλαδή μπορούν αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιήσουν το PowerPoint σε αυτή την ηλικία. Και βλέπουμε ότι οι παιδιά 2-3 ετών χρησιμοποιούν το iPad και το iPhone για να παίξουν παιχνίδια. Γι' αυτό θα ήθελα να ε, ε, δούμε κατά πόσο υπάρχει αυτή η συνδεσιμότητα μεταξύ πολλαπλών χρήσεων που αφορά την προγενέστερη και την ε, τωρινή γενιά. Να γίνεται όμως υπεύθυνη χρήση αυτών των μέσων και ακριβώς αυτό θα πρέπει να λέει και ο καθηγητής, ότι στο διαδίκτυο υπάρχουν καλά και κακά στοιχεία. Υπάρχει η αλήθεια, υπάρχει και το ψεύδος, γι' αυτό θα πρέπει να γίνεται ε, καλή χρήση, σωστή χρήση του διαδικτύου. Να προωθήσουμε την αρχή της επιλεξιμότητας. Στην Πολωνία, στη χώρα μου, σας έλεγα ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στα 7 και 8 τους χρόνια. Ε, πολλές φορές έχουν και μία σάκα τα παιδιά που ζυγίζει πολλά κιλά και πολλές φορές πρέπει να τα βοηθήσω τα παιδιά διότι η σάκα του ζυγίζει πολλά κιλά και πρέπει να τα βοηθήσω στη μεταφορά της σάκας του στο σχολείο. Αυτό λοιπόν που θα μας ενδιέφερε θα ήταν να αποφύγουμε τα βιβλία, τη μεταφορά τους, γιατί θα μπορούσαμε να τα έχουμε σε ηλεκτρονική μορφή. Όχι όλα βέβαια, αλλά πολλά. Μη με παρεξηγήσετε, εγώ προτιμώ το βιβλίο από το iPad, αλλά θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει ηλεκτρονική προσβασιμότητα στα βιβλία, ιδιαίτερα ως προς συγκεκριμένα εγχειρίδια. Δηλαδή, να γίνεται μεγαλύτερη χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων. πολλές φορές είναι ε, πολύ πιο φτηνό να αγοράσει κανείς ένα iPad παρά 50 βιβλία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν πάρα πολλά ε, ερωτήματα που δεν ξέρω καν αν μπορούν να λυθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Μπόρις τώρα ε, έκανε αναφορά στε, εκδοτικά, στους εκδοτικούς οίκους των σχολικών βιβλίων πρόσεξε μην ε, σου κάνουν πρόβλημα από τον εκδοτικό οίκο των σχολικών βιβλίων διότι το ερώτημα για το αν μπορούν να υπάρχουν τα πάντα online είναι αμφιλεγόμενο. Ε, καλό θα ήταν βεβαίως να επιτύχουμε μια ισορροπία μεταξύ των δύο ε, πτυχών. Και γι' αυτό το σκοπό θα χρειαζόμαστε βεβαίως και καθηγητές που θα μπορούν να ανταποκρίνονται σε ένα τέτοιο καθήκον. Και ο χρόνο δεν είναι. Δυστυχώ δεν είναι, δεν είναι όριμη η κατάσταση ακόμη. Πρόσφατα ήμουν σε ένα σχολείο στη, στην ΦΥΡΟΜ, Δεν μπορούσα να καταλάβω. Όλοι είχαν λάπτοπ. Τα ε, παιδιά, ε, εννιάχρονα παιδιά, μπορούσαν με κάποιον τρόπο να μιλήσουν μαζί μου στα ε, αγγλικά. Μπορεί να ήμουν σε ένα πολύ καλό σχολείο βέβαια, αλλά πάντως όλοι οι καθηγητές ήταν εκπαιδευμένοι σε αυτές τις νέες τεχνολογίες και νομίζω ότι χάσαμε πολύ χρόνο ε, έως ότου διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και είμαι σχεδόν βέβαιη ότι στο καινούριο πρόγραμμα Erasmus Plus θα υπάρχουν περισσότερε δυνατότητε για εκπαίδευση και μετεκπαίδευση καθηγητών και γι' αυτόν τον λόγο θα έπρεπε να εξετάσουμε διεξοδικά το πρόγραμμα. Αυτό νομίζω ότι η μετεκπαίδευση καθηγητών είναι ένας από τους στόχους που συμπεριλήφθη και θα ήταν καλό βεβαίως να ε, εστιάσει και ο Ιβάν στην ε, εισηγησή του, στην έκθεσή του, ε, στο τι βοηθητικά εργαλεία υπάρχουν ήδη. Για παράδειγμα, όλοι οι καθηγητές που συμμετέχουν στο e-training του Κομένιους είναι υποχρεωμένοι, ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα στη Στοκχόλμη, ε, και είδα εκεί ήταν 180 καθηγητές οι οποίοι όφυλαν βεβαίως να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες. Πρέπει λοιπόν σε κάθε περίπτωση να εστιάσουμε στην εκπαίδευση των διδασκόντων και μετά να δούμε πόσα χρήματα έχουμε στη διάθεσή μας για να εξοπλίσουμε τα σχολεία. Είναι πολύ δύσκολο για, ε, να, να βρούμε ευρωπαϊκά κονδύλια για τέτοιου είδους υλικό εξοπλισμό. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Το συζητήσαμε και πριν από χρόνια. Είναι πρόβλημα σε ένα πρόγραμμα... Ε, δίνονται χρήματα σε μία χώρα για λάπτοπ, σε άλλη χώρα αυτά δεν αξιοποιούνται. Νομίζω ότι ε, μιλούμε λίγο για έναν τετραγωνισμό της, ε, του κύκλου εδώ πέρα. Ξέρουμε ποιος, ποιος είναι ο στόχος, αλλά να τον επιτύχουμε είναι πολύ δύσκολο. Ε, ίσως από την Κομισιόν ο Ιβάν θα, ίσως η Κομισιόν θα ήθελε να πει κάτι στον Ιβάν. Ε, ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ Καλημέρα σε όλους. Όπως γνωρίζετε η Κομισιόν πρόσφατα ε, υιοθέτησε την πρωτοβουλία Opening Up Education, άνοιγμα εκπαίδευσης, ε, με στόχο κάποιες από τους, ε, ε, να επιτευχθούν κάποιοι από τους στόχους που αναφέρθηκαν εδώ. Πρώτον, έχουμε διαπιστώσει υπάρχει ένα έλλειμμα δεξιοτήτων. Αν δούμε τις θέσεις εργασίας που θα είναι διαθέσιμες σε κάποια χρόνια, θα δούμε ότι σχεδόν όλες οι θέσεις εργασίας, τουλάχιστον 90% θα απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες. Αν όμως δείτε τα αποτελέσματα ΠΙΑΚ που αναφέρθηκαν, μόλις ένας από, τους, ε, από πέντε ε, ενήλικες στην Ευρώπη, θα δείτε ότι ένας ε, στους πέντε δεν έχει τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες ώστε να ανταποκρίνεται σε ένα ε, ε, ψηφιακά προηγμένο περιβάλλον. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ε, θα μπορούσε κανείς να πει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα μεταξύ γενναιών. Οι νέοι ενήλικες μπορούν να ανταποκρίνονται σε, αυτές, τις, σε αυτούς τους στόχους. Η έκθεση ΠΙΑΚ δείχνει ωστόσο ότι παρά το γεγονός ότι οι νέοι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ και μπορούν να κατεβάζουν και να συγκεντρώνουν πολλές πληροφορίες από το ψηφιακό κόσμο. Στην πράξη, όταν αυτές οι δεξιότητες τίθενται σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον, ε, δεν μπορούν οι νέοι να αξιοποιήσουν αυτές τις ικανότητες τους, διότι πολύ συχνά το να βρίσκεται κανείς σε ένα ψηφιακό περιβάλλον δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις δεξιότητες που απαιτούνται σε ένα χώρο εργασίας. Το δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι η αύξηση στη ζήτηση για εκπαίδευση. Θα είναι τεράστια σε παγκόσμιο επίπεδο. Τόσο μεγάλη που κάθε λύση, ε, κάθε λύση που προτείνεται δεν θα καταφέρει να ανταποκριθεί σε αυτή την αύξηση. Σήμερα στον κόσμο έχουμε περίπου 90 εκατομμύρια φοιτητέ ανώτατη εκπαίδευση. Το 2030 ο αριθμό αυτό θα ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια. Άρα ή θα αρχίσουμε να οικοδομούμε πολλά πανεπιστήμια, πολλά τμήματα πανεπιστημιακά ή δεν θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στην ε, αυτή κατάσταση. Και βεβαίως ε, η ψηφιακή εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει τμήμα της λύσης. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι βεβαίως υπάρχει κόστος. Υπάρχει συμπίεση του κόστου, αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι 16 κράτη-μέλη έχουν περιορίσει τους προϋπολογισμούς τους ε, για την εκπαίδευση, για την παιδεία, πολύ πρόσφατα. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και θεωρούμε ότι η ψηφιακή εκπαίδευση μπορεί να έχει μια επίπτωση όσον αφορά την ε, ε, πρόσβαση στη μάθηση ε, λόγω της μείωσης του κόστους. Τέλος, και αυτό αναφέρθηκε ήδη από κάποιο μέλος, είναι ότι η σχέση μεταξύ του καθηγητή και του μαθητή πράγματι αλλάζει. Όταν έχεις πρόσβαση στην πληροφορία και εκτός σχολικής τάξης, οπουδήποτε, τότε ο ρόλος του καθηγητή πρέπει να εξελιχθεί, να γίνει δηλαδή ένας ρόλος που θα διευκολύνει την απόκτηση γνώσεων και να, μην είναι πλέον αυτή η εγκυκλοπαίδεια που ερχόταν ε, κάποτε στην τάξη και απλά ε, έδινε στοιχεία και αριθμούς. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες τάσεις που μας υποχρεώνουν να, να προσεγγίσουμε την τεχνολογία ε, ως ε, εργαλείο για τον εξεχρονισμό. Δεν είναι πανάκια η τεχνολογία για όλα αυτά. Και σίγουρα θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Το να έχει κανείς απλά ένα λάπτοπ στην τάξη δεν θα μας λύσει όλα τα προβλήματα. Αλλά πάντως υπάρχουν πράγματι πολλά πράγματα που μπορεί κανείς να τα επιτύχει μέσω της τεχνολογίας το άνοιγμα της εκπαίδευσης, το opening up education δεν είναι απλά μια έκκληση δηλαδή να ε, θεσπιστούν μέτρα όπως ένα λάπτοπ για κάθε παιδί. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στα σχολεία και στα πανεπιστήμια όπου είναι ενσωματωμένη η νέα τεχνολογία στον τρόπο μάθησης. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο είναι προϋπόθεση αυτό, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και καθηγητές οι οποίοι θα έχουν ψηφιακές δεξιότητες, μάλιστα δεξιότητες υψηλού επίπεδου, υψηλής ποιότητας, να παρέχεται ψηφιακό περιεχόμενο υψηλού υψηλή αξία σε πολλέ γνώσει. Υπάρχουν λοιπόν πολλέ προποθέσει για να επιτύχουμε του στόχου μα. Ε, το Opening Up Education τονίζει τρει βασικού τομεί και αυτοί οι τρει τομεί ανταποκρίνονται και στην οργάνωση, στο ε, στην οργάνωση της εκπαίδευσης αφορά αφενός την εκπαίδευση των καθηγητών αλλά αφορά επίσης την ε, υποστήριξη προς ε, τα ιδρύματα που θα ήθελαν να αναθεωρήσουν τα οργανωτικά τους μοντέλα ώστε να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα της επαλήθεσης και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων. Το δεύτερο στοιχείο είναι η προώθηση ε, ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από αυτή την άποψη μία από τις κοινοτομίε που εισάγει το Erasmus Plus που μόλις ε, υπερψηφίσατε σήμερα το πρωί είναι η δέσμευσή μας όλο το εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus Plus να ε, είναι δημόσια προσβάσιο, προσβάσιμο και να χαρακτηρίζεται από ανοιχτέ άδειε χρήση. και τρίτο ζήτημα η συνδεσιμότητα διότι χωρίς σύνδεση δεν μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Το Opening Up Education είναι ε, πρωτοβουλία της Επιτρόπου ε, Βασιλείου και της Αντιπροέδρου Νελικρούς και στόχος μας είναι να συνδυάσουμε την παιδεία με τις νέες τεχνολογίες. Ε, προσδιορίσαμε 23 δράσεις. Όπως είπα δεν πρόκειται να είναι πανάκια που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα προβλήματα, όμως έχουμε προσδιορίσει αυτές τις 23 δράσεις, τις έχουμε συζητήσει ε, ε, με τους ενδιαφερόμενους σε μια ευρεία διαβούλευση για χρόνο μεγαλύτερο του ενός έτους και νομίζουμε ότι είναι τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε τώρα προκειμένου να κάνουμε βήματα μπροστά στον τομέα αυτό. Ενδεχομένως σε κάποια χρόνια θα ανακύψουν καινούργια ζητήματα, άλλα ζητήματα από αυτά που, ε, άλλα από αυτά που συζητούμε σήμερα, αλλά θεωρούμε ότι αυτά που προτείνουμε για το Opening Up Education είναι αυτή τη στιγμή ρεαλιστικά, μπορούν να χρηματοδοτηθούν με το πρόγραμμα Erasmus Plus, αλλά και με τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση με ορίζοντα τον 2020. Δεν πρόκειται για νέα χρήματα, αλλά πάντως τονίζουμε κάποιες νέες πτυχές που τα προγράμματα αυτά θα μπορούν να υποστηρίξουν σε αυτήν την ε, νέα ε, φάση χρηματοδότησης. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Πολύ χρήσιμα και για τον Ιβάν. Ιβάν, θα ήθελες να πεις κάτι? Όχι τότε μπορούμε να ψηφίσουμε για την έκθεσή σου τον Δεκέμβριο. Ναι, το, το σχέδιο θα μας το παρουσιάσεις τον Δεκέμβριο και η ψηφοφορία θα γίνει το Φεβρουάριο. Δεν είναι πήγον, θα είναι μάλλον από μία από τις τελευταίες ψηφοφορίες μας. Ευχαριστώ κύριε Φερέιρα. 10. Έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών. Πήρατε το email. Ε, διάφορα, δεν υπάρχει κάτι. 12. Να ευχαριστήσω τους ε, διερμηνείς, ευχαριστώ πολύ όλους εσάς στις καμπίνες και ξανασυναντιόμαστε η επόμενη συνεδρία 27 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Είναι η ολοήμερη συνεδρία μας εκείνη τη μέρα 27 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ. Γεια σας.